So, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, ώρα είναι 3 και 3, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε μπροστά σας την ημερήσια διάταξη, υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι, άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών ε, για την ε, Συμφωνία Ελευθέρωσης Αλλαγών με το Βιετνάμ. Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι λόγω του ότι το πιθανότερο είναι να μην ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι το τέλος της θητείας, θα αναβάλουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ε, για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ και την έκθεση IPA. Ο εισηγητή συνεχίζει τι προσπάθειέ του και εάν τα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό εντό τη θητεία αυτή και να έχουμε υπογραφή δηλαδή από το Συμβούλιο σύντομα, διότι άκουσα ότι η Σεσίλια Μάλμστρομ είναι διατεθειμένη να πάει στο Ανόη, θα θέσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες. Ωραία. Έχουμε μαζί μας δύο προσκεκλημένους, την Αράντσα Γκονζάλες και τον ε, πρέσβη μας ε, στον ΠΟΕ, τον κύριο Νόικλε. Και το θέμα που έχουμε είναι η κατάσταση των κοινών πρωτοβουλειών ε, ένα έτος μετά την 11η Υπουργική Συνδιάσκεψη. Η διάσκεψη αυτή ήταν απογοητευτική. Οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικές προσεγγίσει όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, θέματα των δύο φύλων κλπ. Δεν καταφέραμε όμως να πετύχουμε συμφωνία σε κανένα από αυτά τα θέματα, ούτε καν στις ενισχύσεις για την αλλήλεια, που θεωρούσα ότι είναι από τα πιο εύκολα θέματα και που συνδέεται και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι, ο ΠΟΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα είχαν κάποια επιτυχία. Ο ΠΟΕ υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Τέλος πάντων, έτσι έχει η κατάσταση. Και μπορούμε να συζητήσουμε τώρα το θέμα αυτό με τους δύο πυρογνώμονές μας. Δίνω το λόγο πρώτα στην Αράντσα Γκονζάλες. Παρακαλώ. Thank you very much, Bern. Thank you for the invitation to come to the European Parliament. It's about the year since Buenos Aires took place. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας χρόνος πέρασε περίπου από την ε, συνάντηση ε, στο Buenos Aires. Ε, είναι σωστό και χρήσιμο να δούμε τι ακριβώς συνέβη από την Υπουργική Συνάντηση στην Αστάνα. Νομίζω το Buenos Aires ήταν σημαντικό στο πλαίσιο αυτών των εμπορικών εντάσεων που βιώνουμε διότι δεν εστιαστήκε μόνο στο άνοιγμα του εμπορίου, αλλά στο δίκαιο και βιώσιμο και συμμετοχικό εμπόριο. Πρόκειται για μια δουλειά που συνεχίζεται. Το πρόγραμμα ήταν πιο σημαντικό από τα παραδοτέα που έχουμε μέχρι σήμερα. Αλλά η κατεύθυνση είναι σωστή. πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να έρωμε εμπόδια προς το διεθνές εμπόριο. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που θα βοηθάει στην συμμετοχικότητα, στην συμπεριληπτικότητα μάλλον και στη βιωσιμότητα. Πρέπει να έχουμε πιο συμπεριληπτικό εμπόριο, πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις γυναίκες στο στον τομέα του εμπορίου. Δεν θα μπω στα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα το κάνει ο Μάρκ. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λοιπόν. Εδώ δεν μιλούμε τόσο στην δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το να καλύψουμε περιοχές, παιδεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για αυτές και ένα από αυτά είναι η πιο εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν σχέση με το εμπορικό επιχειρήν. Στον ΠΟΕ έχουμε εκινήσει μία διαδικτυακή πύλη helpmetrade.org που είναι δωρεάν και προσβάσιμη για όλους και όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες της αγοράς, σε market intelligence. Θα αυξηθεί, θα προσθέσουμε στον όγκο των πληροφοριών που ήδη έχει η πύλη αυτή. Δεν προσπαθούμε να επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά να συγκεντρώσουμε την πληροφορία που έχουμε σε ένα σημείο. Για τις γυναίκες στον εμπορικό τομέα, να θυμίσω γιατί είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι δεν θυμόμαστε ή δεν κατανοούμε γιατί πρέπει να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Ο λόγος είναι ότι έτσι εξασφαλίζουμε περισσότερη μεγέθυνση οικονομική και καλύτερης ποιότητας. Μόνο ένα στους πέντε εξαγωγείς σήμερα είναι γυναίκες. Ένας εξαγωγέας που ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι γυναίκα παράγει περισσότερες θέσεις για γυναίκες Γιατί έχουμε στατιστικά στοιχεία που συγκρίνουν τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες με εκείνες που διευθύνονται από άντρες και έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας κατά μέρο Κατά μέσον όρο επίσης έχουμε 1,6 φορές καλύτερο μισθό κατά μέσον όρο που καταβάλουν, που πληρώνουν οι επιχειρήσει αυτέ. Είναι λοιπόν σημαντικό να προχωρήσουμε στην συμμετοχή των γυναικών στο διεθνέ εμπόριο. Τι έγινε τώρα από την διακήρυξη του Buenos Aires. Ανταλλάσσουμε εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές, μεθοδολογία. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε για να άρρωμε τα εμπόδια για το εμπόριο των γυναικών. Και έκτοτε έχουμε τρεις νέους συνυπογράφοντες. Είχαμε διοργανώσει τρεις εκδηλώσεις γνώσης για την ανάλυση των δημοσίων προμηθειών της ε, αλυσίδας αξίας για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επί των οποίων θεματικών συλλέγουμε γνώση από όλο τον κόσμο που και θα συντάξουμε από αυτού και ένα εγχειρίδιο για την επόμενη υπουργική. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι και άλλοι φορείς η ΠΕΚ, η Προεδρία η Χιλιανή φέτος, για παράδειγμα, τοποθέτησε το θέμα την διάταξή της. Η Ιαπωνία επίσης το έπραξε. Έχουμε και πέντε μελέτες πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Γκάμπια και το έχουν συζητήσει το θέμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Νεπάλ, το Μαυροβούνιο και άλλες χώρες. Στη διαπραγμάτευση λοιπόν των εμπορικών συμφωνιών, των συμφωνιών ελευθερών συναλλαγών, υπάρχουν όλο και περισσότερα κεφάλαια για την ισότητα των φύλων και για τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών. Εμείς είμαστε ένας συνεργάτης και εταίρος της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να διεξαγάγουμε έρευνες σε 12 κράτη-μέλη για να δούμε μη δεσμολογικά εμπόδια μέσω του θεματολογίου του φύλου. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια εμπόδια προς τις γυναίκες. Έχουν αντίκτυπο. Και άλλη μια περιοχή από τις οποίες συνεργαζόμαστε μαζί σας είναι για να αναπτύξουμε ένα εργαλείο το οποίο θα ονομάζεται Sea Trades Outlook, λέει ο Μιλήτρια, για να δούμε πόσο φιλικό είναι το περιβάλλον μιας συγκεκριμένη χώρας προς τις γυναίκες, προς το γυναικείο εμπόριο. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια και νομίζω ότι το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε για την επόμενη υπουργική διάσκεψη είναι επί τη βάση της ε, αναφοράς που υπευλήθη στους υπουργού, πώς μπορεί το θέμα αυτό να είναι όλο και πιο συστηματικά μέρος της δουλειά του ΠΟΕ, όχι ως δουλειά του περιθωρίου, αλλά πώς θα ενταχθεί στο βασικό του πρόγραμμα. Και με αυτά, Πρόεδρε, ολοκληρώνω την σύντομη εισήγησή μου των όσων συνέβησαν από τον Thanks a Ελία, σας ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο τον κύριο Πρέσβη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε η Αράντσα λέγοντας το εξή. Πώς έχουν τα πράγματα τώρα σε σχέση με τις τρεις άλλες κοινέ πρωτοβουλίες οι οποίες ζήτηκαν στον Buenos και τέθηκαν σε εκείνης. Όπως είπατε πρόεδρε, στον Buenos ήταν απογοητευτικό να αφορά τα αποτελέσματα. Ε, δέθηκαν όμω σε οι κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες λειτουργήσαν το 2018, θα συνεχιστούν το 2019 και αρχίζουμε τώρα να βλέπουμε τα πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτές οι τρεις άλλες κοινέ πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν σχέση με το ε, ηλεκτρονικό εμπόριο, με την ε, δήλωση για τις ε, ΜΜΕ και για τα θέματα που αφορούν τις επενδύσεις και την διευκόλυνσή τους για θέματα ανάπτυξης. Κάποια μέλη, 60 ή 70 σε σύνολο στο Buenos Aires, άρχισαν διερευνητικές ομιλίες Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στα πλαίσια του ΠΟΕ. Οι συζητήσεις αυτές ήταν αρκετά εντατικές το 2018 και τέθηκαν οι βάσεις ώστε να τεθεί το γενικότερο ερώτημα. Δεν θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε περισσότερο και να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για όλα αυτά τα θέματα τα εμπορικά που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πριν από δύο εβδομάδες, στον Ταβός, σε μία μήνυ υπουργική διάσκεψη, 50, ε, συγγνώμη, 70 περίπου από τα μέλη, ε, περίπου 70, επαναλαμβάνω, άρχισαν σιγά σιγά τις διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις της 6η ε, Μαρτίου επισήμως που θα έχουμε την πρώτη μας συνεδρίαση. Σε σχέση με τους ε, αρχικά μέλη τα οποία άρχισαν αυτές τις συζητήσεις στο Buenos Aires, πρέπει να πω ότι αυξάνονται τα μέλη τα οποία προσυπογράφουν και προχωρούν. Ένα πολύ σημαντικό μέλος είναι η Κίνα δεν είχε υπογράψει την κοινή πρωτοβουλία εκείνη, αλλά τώρα μπήκε και εκείνη στο άρμα των διαπραγματεύσεων μετά από τη Βραζιλία. Έχουμε λοιπόν πολλά μέλη, όπως σας λέω, που εκπροσωπούν περισσότερο από 90% του παγκοσμίου εμπορίου και που θα αρχίσουν αυτές τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν ακόμη και κάποιοι πολύ σημαντικοί απόντες, θα έλεγα την βία, η Νότιος Αφρική και μεγάλο μέρος των κρατών της Αφρικής. Αλλά η κοινή πρωτοβουλία αυτή για το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να πω ότι προχώρησε πολύ υπό την ηγεσία της Σιγκαπούρης, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και όπως ήδη είπα θα αρχίσουμε πραγματικά τις διαπραγματεύσεις στις 6 Μαρτίου. Η δεύτερη κοινή πρωτοβουλία που ήταν επίσης πολυμερούς ε, φύσης, ήταν ε, ε, αυτή που αφορούσε την δημιουργία ενός πολυμερούς πλαισίου για την διευκόλυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη. Η ιδέα δεν είναι να μπούμε μέσα στους σκληρούς κανόνες των επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συνειδητοποιούμε απολύτως. Δεν ε, θέλουμε να μπούμε σε τέτοιες λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα, αλλά να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για επενδυτικούς λόγους, για, με για αναπτυξιακούς λόγους. Και έτσι Είμαστε στην εξή φάση. Έχουμε ένα checklist, έναν ε, κατάλογο των ε, πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της, ε, του πολυμερούς αυτού πλαισίου διευκόλυνση των επενδύσεων. Το επόμενο εξάμεινο θα συζητηθούν αυτά τα θέματα βάσει των υπαρχόντων παραδειγμάτων και των βελτίστων πρακτικών και η ιδέα είναι μετά να προχωρήσουμε τον Ιούνιο το 2020 στην συνεδρία της Αστάνα, όπου θα φτάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση αυτού του πολυμερούς πλαίσιου. Τώρα, το τελευταίο θέμα. Στις υπηρεσίες οι, ε, οι κανονισμοί που θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε χώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο άρχισε ήδη από το γύρο των συνομιλιών της Ουρουγουάης, μετά που ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις στα πλαίσια του ΚΑΤ, είπαμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε όσον αφορά αυτό το θέμα, δηλαδή τους κανόνες που αφορούν τις εξαισιοδοτήσεις, τις άδειες αυτών οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες σε κάθε χώρα. Αναλώσαμε πολλά χρόνια σε συζητήσεις επί αυτών των θεμάτων. Αλλά Πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα πολυμερή, δεδομένου ότι όλα αυτά τα θέματα άπτονται και άλλων πολύ σημαντικών που, έχουν παρεμφερεί, που είναι παρεμφερεί. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει ε, να μπούμε σε άκαμπτους κανόνες, διότι θα πρέπει να αφήσουμε χώρο ώστε ο καθένας να μπορέσει σωστά να αναπτύξει την πολιτική του. Είπαμε ότι θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα κείμενο στο οποίο θα περιέχονται όλα αυτά τα βασικά θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια των υπηρεσιών αυτών και των κανόνων που πρέπει να ισχύουν. Τώρα έχουμε για τις ε, υπηρεσίες επίπεδο περίπου ένα καλό κείμενο, περίπου 65 με 70 μέλη είπαν ότι πραγματικά τα ικανοποιεί το κείμενο αυτό. Υπάρχουν κάποια ε, δευτερευώσει σημασία θέματα πρέπει να επιληθούν. Και το δεύτερο θέμα είναι τι κάνουμε τώρα με αυτό το κείμενο. Όταν θα ολοκληρωθεί, πώς θα προχωρήσουμε. Θα, έχουμε, θα θέλουμε να έχουμε ένα κείμενο που να ισχύει ε, διεθνώς ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται από μέλη του ΠΟΕ, ξέροντας ότι κάποια κράτη-μέλη κατηγορηματικά μέχρι τώρα το απορρίπτουν, κάτι τέτοιο. Ή σιγά σιγά θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία κάθε χώρα χωριστά θα μπορεί να αναλάβει, να αναλαμβάνει τέτοιου είδους δεσμέσεις ε, σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ. Άρα Αυτά είναι τα θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούμε τις επόμενες εβδομάδες για να δούμε τι γίνεται τελικά με το θέμα αυτό, ποια θα είναι η κατάληξη όλου αυτού του φακέλου και αν θα προχωρήσουμε ε, έτσι όπως είμαστε τώρα ή θα έχουμε ε, αποτελέσματα τα οποία θα εφαρμοστούν διεθνώς. Στο Buenos Aires τώρα είπαμε ότι θα πρέπει για τα θέματα ε, που αφορούν ε, την ε, αλληλεία και διάφορες σχετικά θέματα να προχωρήσουμε ή θα τα αφήσουμε έτσι. Θέλουμε, όπως ελέγχθηκε στην μήνυ υπουργική συνεδρίαση στον Ταβό να προχωρήσουμε έτσι, αλλά θέλουμε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στον τομέα αυτό μέχρι το τέλος του 19. Πριν από την Αστάνα, λοιπόν, θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, δεδομένου ότι μέχρι το 2020, όπως συμφώνησα και οι Υπουργοί, θα πρέπει να έχουμε ένα σχετικό κείμενο. Θέλουμε λοιπόν μέχρι το τέλος του 2019 να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας και να έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις δεδομένου ότι θέλουμε η MC να μπορέσει στα πλαίσια της εφόρου ανάπτυξης να δώσει ισχυρά μηνύματα ακόμη και σε θέματα που αφορούν την ενέργεια. Σας ευχαριστώ. ευχαριστώ. Υπάρχουν Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Υπάρχουν ερωτήσεις. Uh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη, που μας ενημερώσατε σχετικά με διάφορες πτυχές των εργασιών εντός του ΠΟΕ. Το ενδιαφέρον δεν αντικατοπτρίζεται από την παρουσία του στην αίθουσα. Ε, ε, μας ενδιαφέρουν πολύ τα θέματα του ΠΟΕ και οι πολιτικές ομάδες ασχολούνται με το θέμα αυτό και η δική μου πολιτική ομάδα είναι υπέρ του να διατηρηθούν οι προσπάθειες για ε, ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος που να αντικατοπτρίζει την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα στα κράτη-μέλη του ΠΟΕ. Αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο αναφορά μα. Και όπω είπατε, κύριε Πρέσβη, η στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη ε, είναι ένα από αυτά τα σημεία αναφορά και αναφερθήκατε στο σημείο 14.6 ω ε, συγκεκριμένη παρέκκληση. Θα πρέπει να Προσπαθούμε πάντα να εφαρμόζουμε οριζόντια τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να ε, ξεπεράσουμε την ε, φτώχεια, για παράδειγμα, να λύσουμε το πρόβλημα της φτώχειας. Υπάρχει και το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όταν ε, δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας, συμφωνήθηκε και στον Ταβός ότι θα πρέπει να δοθεί νέα ορμή στο θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. στο Δεβόσε συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε περισσότερο εις βάθος. Ε, η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με την Συμφωνία Διευκόλυνσης Εμπορίου και με την ε, Συμφωνία Διευκόλυνσης των Επενδύσεων. Στην πράξη, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε οι οικονομίες των φτωχότερων χωρών, να τις ονομάσω έτσι, θα μπορούν να αποτελέσουν τέρο στις επενδύσεις και να μην χρησιμοποιούνται μόνο ως χώρος για πραγματοποίηση των στόχων των επενδυτών. Δηλαδή, στην ε, παγκόσμια αλυσίδα αξίας, πώς μπορούν να ενσωματωθούν οι χώρες αυτές, ώστε να μην υποκύπτουν στην οικονομική ισχύ των μεγάλων χωρών. Τρίτη ερώτηση. Δεν αναφέρατε την συζήτηση για μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το που βρισκόμαστε και δεδομένου του παγκοσμίου εμπορίου και των ε, συγκρούσεων που βλέπουμε ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, για παράδειγμα, και άλλες χώρες. Ευχαριστώ κυρία Όταλα, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για τις προσπάθειές σας να θέσετε πάλι στο επίκεντρο το πολυμερές σύστημα εμπορίου. Ιδιαίτερα χάρηκα που άκουσα ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Η εργασία σας εδώ και πολλά χρόνια είναι πολύ χρήσιμες ε, στον τομέα αυτών. Η ερώτησή μου ε, συνδέεται με την ερώτηση του συναδέρφου Σόλς, διότι και μετά τον Buenos Aires είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα πια προσπαθεί να θέσει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση. Αυτό είναι κάτι που αφορά τις εργασίες σας, διότι νομίζω ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι έχουν να παίξουν ρόλο στην εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Το ε, σχέδιο δράσης για τον βιώσιμο χρηματοοικονομικό τομέα, το θέμα της ε, ταξονομίας όπως ονομάζεται, ε, έχει να κάνει με την ε, εκπόνηση των κριτηρίων για τον βιώσιμο χρηματοοικονομικό τομέα. Πώς αντικατοπτρίζονται αυτά στις δικές σας εργασίες. Ε, σας ευχαριστώ και... Ε, και θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, και... Ε, όσον αφορά τις έξι προσεγγίσεις, ε, υπάρχει συνένεση ε, μεταξύ πολλών κρατών όχι ωστόσο και των 164. Θέλουμε να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα με το οποίο να συμφωνούν όλοι, ώστε τελικά ο ΠΟΕ να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο πολυμερών διαπραγματεύσεων, στο οποίο να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Πρόκειται λοιπόν για ένα μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σχετικά με τη νέα προσέγγιση εντός του ΠΟΕ. Δεύτερον, ε, τι γίνεται με το γύρο της Δόχα. Ένας μεγάλος εταίρος, ε, είχαμε τη συζήτηση για την Ινδία στη διευθύνουσα ομάδα. Λέει ότι η Ινδία λοιπόν λέει ότι δεν θα κάνει τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα. Πώς ε, θα αντιμετωπίσετε εσείς ε, αυτό το μήνυμα. Και τρίτον, δεν αναφερθήκατε στο θέμα του δευτεροβάθμιου διοικητικού οργάνου. Έχουμε κάποιες προτάσεις ε, της Αφρικανικής Ένωσης, του Καναδά, έχουμε κάποιες επικρίσεις από τις Ηνωμένε Πολιτείες, έχουμε απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τι ακριβώς γίνεται λοιπόν και πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη γενικότερη συζήτηση. Ο κύριος Ρούμπιχ επίσης έχει μια ερώτηση να σας θέσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη αλλά δεν είναι πολύ εύκολες ε, οι αερομεταφορές ε, στις μέρες μας. Ε, είναι μια διασυνοριακή υπηρεσία και όταν απεργεί ένα αεροδρόμιο, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν όλοι να καταφτάσουν στην ώρα τους. Χαιρόμαστε όμως που καταφέρατε να έρθετε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Buenos Aires ήταν εκτενής οι διαπραγματεύσεις και γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να συμφωνήσουν τελικά όλοι οι εταίροι. Πολύ συχνά τα ατομικά συμφέροντα πρέπει να τεθούν κατά μέρος προς όφελος των κοινών συμφερόντων. Θέλουμε ένα σύστημα πολυμερές που να βασίζεται στους, σε κανόνες. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για την οικοδόμηση δυναμικού, το capacity building, να μιλήσουμε για τα ισχυρά ε, σημεία του ε, ΠΟΕ. Ο Τραμπ ε, έχει καλέσει τις ε, χώρες του ΝΑΤΟ να επενδύουν το 2% του ΑΕΠ τους σε εξοπλισμούς. Ίσως ε, δεν θα λέγω ότι συμφωνώ με αυτό, αλλά μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε αν το σύστημα υπό την παρούσα του μορφή, όπως αναφέρθηκε και στο Buenos Aires, ε, να απαιτεί επιγόντως ε, μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει από τη μία μεριά το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους υπουργούς δηλαδή, από την άλλη έχει ένα κοινοβούλιο όπου εκπροσωπείται και η αντιπολίτευση. Και ακριβώς αυτό είναι και το ισχυρό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως θα πρέπει να έχουμε κάτι παρόμοιο στον ΠΟΕ. Στις, βιομηχανικές χώρες αλλά και στις λιγότερο αναπτυσμένες χώρες ε, είναι απαραίτητο νομίζω είναι καλύτερο ε, να δοθούν ε, όλες να αντιπροσωπεύονται όλες οι απόψεις απέναντι στο κοινό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται 28 κράτη-μέλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ένα παρόμοιο σύστημα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ο ΠΟΕ αυτή τη στιγμή έχει 640 υπαλλήλους με προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ. και ο πρόεδρος μας ε, πολύ σωστά επισήμανε ότι ίσως ε, θα είναι χρήσιμο να αυξήσουμε τους πόρους, διότι αν συγκρίνουμε το δευτεροβάθμιο δικαιωτικό όργανο ε, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν διαφορές και όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. Ε, η υπουργική διάσκεψη, η συνέλευση, ε, ο ΠΟΕ αυτός καθ' αυτός, ε, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, όλα αυτά είναι χρήσιμα όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά τα έχει καταφέρει με αυτό το τετράπτυχο. Ρωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να έχουμε μια επίσημη κοινοβουλευτική συνέλευση στον ΠΟΕ. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, θα ήταν δυνατόν να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να έχουμε και στον ΠΟΕ αυτόν τον συμβουλευτικό χαρακτήρα. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τι θα καταφέρουμε μέχρι το 2020, την 12η Υπουργική Διάσκεψη δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ, Αράντσα. Helmut Scholz. Uh, it is indeed... Πράγματι, είναι η στό, οι στόχοι της ε, βιώσιμης ανάπτυξης που πρέπει να κοιτούμε, αν και πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο για την διεθνή εμπορική κοινότητα να συσχετιστεί με αυτούς τους στόχους. Από την άλλη μεριά αυτοί οι στόχοι καμιά φορά δεν συνδέονται απόλυτα με το διεθνές εμπόριο με τον καλύτερο τρόπο. Εν πάση με το υπαριθμό 17 των SDG λέμε ξεκάθαρα, αναφερόμαστε μάλλον στο, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ε, βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση, στην ε, εκρίζωση της ένδειας και είναι καθρέφτης ε, της συμφωνίας του ΠΟΕ στο προήμιο. Είναι καλό δηλαδή να αλλάξουμε, αν θέλετε, την κατεύθυνση και των δύο πλευρών για να συσχετίζονται καλύτερα. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουμε τεράστια ε, δυναμικό εδώ και χωρίς να σκεφτόμαστε απλώς το B2B αλλά και το B2C, δηλαδή τη σχέση με τους καταναλωτές που πάρα πολλοί φορείς μικρής κλίμακας σε πολλές χώρες μπορούν να πραγματοποιήσουν. Επομένως, αφενός είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι οι διαπραγματεύσει στον ΠΟΕ θα είναι όσο πιο πλήρης γίνεται, γιατί έχουμε ευκαιρία για πρώτη φορά να ρυθμίσουμε μια περιοχή ε, που αφορά στο διεθνές εμπόριο και με όλους συμμετέχοντες στο τραπέζι. Δεύτερον, σημαντικό και περισσότερο για τα ευρωπαϊκά θέματα, καθότι ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα συμμόρφωσης ε, εντός του εδαφούς τους, θα πρέπει να λάβετε και υπόψη σας τις ευκαιρίες και το αυξανόμενο κόστος που αντιμετωπίζουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για τις διευκολύνσεις, αυτό που κάνουμε στο Διεθνές Κέντρο είναι να συνεργαζόμαστε με μεγάλο αριθμό χωρών για να τις βοηθούμε να κατανοούν πόσο μπορούν, πώς μπορούν καλύτερα να προσελκύσουν ποιοτικές επενδύσεις με καλύτερη χαρτογράφηση αλλά εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι, έχουμε, ότι πρέπει να γίνει καλύτερη δουλειά με τις αναπτυσσόμενε χώρες. Υπό τη συμφωνία του ΠΟΕ αυτό θα γινόταν πιο εύκολο, αλλά δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανάπτυξη του δυναμικού μιας χώρας, ώστε να, έχουμε, να αναπτύσσει η χώρα αυτή επενδυτικά έργα που θα προσελκύουν ποιοτικού επενδυτές. Για την βιώσιμη χρηματοδότηση μπορείτε να σημειώσετε ότι στην επόμενη αναθεώρηση της ε, ετήσιας έκθεσής μας για το θέμα αυτό εστιαζόμαστε στη χρηματοδότηση της βάσης της πυραμίδας. Δηλαδή με πιο απλούς όρους πώς μπορούμε να φέρουμε το μεγάλο κεφάλαιο στις μικρές επιχειρήσεις. έχουμε εστιαστεί ήδη αρκετά στις υποδομές, αλλά όχι τόσο στην καλύτερη χρηματοδότηση, περισσότερη χρηματοδότηση και οικοδόμηση των αγορών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν οικοδομηθεί, υπό την οπτική, υπό το πρίσμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και τα ευρωπαϊκά σχέδια, τα επενδυτικά, ιδιαίτερα το αφραγανικό, είναι ένα πολύ καλό χρήσιμο πεδίο ώστε να προσελκυθεί κεφάλαιο στη βάση της πυραμίδας. Τώρα, είναι αλήθεια ότι κινούμαστε προς ένα πιο ευέλικτο σύστημα. Για μένα το θέμα δεν είναι το είδος της πολυμέρειας, αλλά αν είναι ανοιχτό ή κλειστό. Αν καλύπτουμε το 95% του διεθνούς εμπορίου και αυτό το κάνουμε με τρόπο ανοιχτό και διαφανή, επιτρέποντας σε όλους να κατανοήσουν, να καταλάβουν τους νέους κανόνες, δεν θα θεωρούσα ότι κατακαιρματίζουμε το σύστημα. Τώρα, άλλο θέμα είναι να το κάνει κανείς αυτό στη γωνιά του, για τον εαυτό του, για λογαριασμό του. Επομένως, είναι το είδος της πολυμέρειας και όχι η ονοματολογική διαφορά μεταξύ multilateralism και plurilateralism που έχει σημασία. Επομένως είναι πιο αποτελεσματικό αυτό να συζητηθεί εντό του ΠΟΕ παρά εκτό. Τώρα για την κοινοβουλευτική συνδάσκεψη τα κοινοβούλια έχουν ρόλο να διαραματίσουν το Διεθνέ εμπόριο. Το έχουμε δει αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε μικρότερο ρόλο παλαιότερα και σήμερα έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι πρέπει να προσελκύσει, να αυξήσει την νομιμότητα, την νομιμοποίηση της όλης ε, διαδικασίας. Η συνδιάσκεψη θα έπρεπε να είναι για όλα τα μέλη. Η IPU δυστυχώς δεν είναι για όλα αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα ήταν ένα, μια πολύ καλή κατεύθυνση για να αυξήσουμε και την νομιμότητα αλλά και την ποιότητα της συζήτησης. Δεν ξέρω κατά πόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην επίλυση διαφορών, όπως και δεν διαδραματίζει υπό το πλαίσιο του δικαστηρίου. Αυτό είναι βεβαίως η προσωπική μου τοποθέτηση, Πρόεδρε. Thank you. Let me... Uh, uh, Ο κύριος Πρέσβης, σας ευχαριστώ. επί των πτυχών που η Αράντσα ίσως δεν κάλυψε τόσο αναλυτικά και παρότι βέβαια μπορούμε να μιλούμε πολύ ώρα για όλα αυτά, για την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι ένα θέμα που είναι επιτάπητος στον ΠΟΕ και το θέμα γίνεται όλο και σημαντικό. Είναι επίση αλήθεια ότι μέχρι τώρα Ως προς τον επιχειρησιακό αντίκτυπο, το θέμα αυτό υπήρξε μικρής κλίμακας. Ο μόνος σημαντικός φάκελος στο τραπέζι που συσχετίζει μεταξύ της δημιουργίας των κανόνων του ΠΟΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η αλληλεία. Υπάρχουν και άλλες θεματικές, το εμπόριο σε γεωργικά προϊόντα, σε ενισχύσεις για ορυκτά καύσιμα, στην κλιματική αλλαγή, αυτές οι θεματικές αναφέρονται όλο και περισσότερο. Και είναι σημαντικό να σημειώσει κανείς ότι στην πολυμερή διάσταση του διαλόγου για τα θέματα αυτά, η υπερβολική διάσταση έχει υπογραμμιστεί πολύ περισσότερο από την κοινωνική διάσταση, η οποία είναι πολύ σημαντική στις διμερείς επαφές της Ένωσης με τους εταίρους της μέσω FTA, αλλά στην Γενέβη ο σχετισμός μεταξύ εμπορίου και απασχόλησης ή εμπορίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ακόμα ελλειπής. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα δούμε το περίγραμμα λέει ο του αποτελέσματος που θα προκύψει Τώρα ε, είχαμε μια προσέγγιση όπου όλοι θα μπορούσαν να προσθέσουν, να συνεισφέρουν τη δική θεματική και τώρα έχουμε ένα μακρύ κατάλογο θεμάτων. Θα δούμε τι τελικώς θα συμπεριληφθεί στο κείμενο. Και η πολιτική πρόκληση εκεί θα είναι να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία που θα συμπεριλαμβάνει όσο το, όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Μια ευέλικτη δομή που θα λέει ότι μάλλον το να απαιτήσουμε ότι όλοι θα κάνουν εξίσου σε όλες τις θεματικές μάλλον δεν είναι τόσο ρεαλιστικό. Για τις διευκολύνσεις επενδύσεων, όπως είπα και στην εισαγωγή, εδώ το σκεπτικό δεν είναι η προστασία ή η πρόσβαση στην αγορά, η προστασία των επενδύσεων ή η πρόσβαση στην αγορά, αλλά πώς τα μέλη μέσω καλών πρακτικών, μέσω της διαφάνειας, μέσω ενιαίας στηρίδας στην οποία θα μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα οι επενδυτέ, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα, ένα περιβάλλον φιλικό προς του επενδυτέ και που θα του προσελκύει. Αλλά δεν έχουμε κατά νου να επιβάλλουμε κανόνες σε κανένα μέλος. Να έχουμε απλώς έναν οδηγό, αν θέλετε, μια συλλογή καλών πρακτικών για τις επενδύσεις. Ώστε να τις προσελκύουμε περισσότερο πολύ σημαντικό θέμα στο οποίο δεν αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου, γιατί θεώρησα ότι έπρεπε να εστιαστώ στις κοινέ πρωτοβουλίες του Μπίνος Άρες, ήταν πολύ σημαντικό θέμα η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ. Να σας πω ένα-δύο πράγματα σχετικά. Οι τρεις πυλώνες του οικοδομήματος του ΠΟΕ απαιτούν μια επανεξέταση, μια μεταρρύθμιση οι κοινοί κανόνες, η υλοποίηση των υφισταμένων, οι πληροφορίε που χρειάζονται σχετικά με αυτό και τρίτον η επίλυση διαφόρων. Για το τελευταίο γνωρίζετε την κατάσταση, το ρολόι τρέχει, ο χρόνος τρέχει. Θα έχουμε μόνο ένα μέλος στο, ε, στον φορέα εφέσεων και μετά θα φτάσουμε σε ένα μπλοκάρισμα και κανείς δεν ε, υποβάλλει πρακτικές προτάσεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο μαζί με άλλους εννέα εταίρους έχουν υποβάλει πρόταση και τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία από ότι πριν από αυτή την πρόταση. Το 18 στο υψηλότερο, στο υψηλότερο επίπεδο σώμα του προεπέραν του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι το Γενικό Συμβούλιο συζητήσαμε μία άτυπη διαδικασία υπό την οποία οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων θα συζητηθούν. Και η πρώτη συνάντηση που θα γίνει από αυτού είναι μεθαύριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν, έχουν δηλώσει και θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα θέματα τα οποία έδειξαν οι Αμερικανοί για να δούμε τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει και τι μπορούμε, πώς μπορούμε να υποκαταστήσουμε τα, τα σημεία που θεωρούν αρνητικά. Γιατί προς το παρόν ε, είναι κάπως αυτιστική η στάση τους των Αμερικανών. Λένε ότι οι φορείς του σώματος εφέσεων θα πρέπει να μείνουν στους κανόνες του 96 και να είναι καλά παιδιά. Εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα προκύπτει από τη διευκρίνηση που απαιτείται για αρκετούς κανόνες σχετικά με την επίλυση διαφορών και εξού και η πρόταση που υπευλήθη. Για την ερώτηση του κυρίου Λάγκε για τις κοινέ πρωτοβουλίες, πλησιάζουμε σιγά σιγά στην ολοκλήρωση, στον τερματισμό του single undertaking. Αύριο και θα συνεχίσουμε την συζήτηση για τα γεωργικά θέματα που είναι τα κυρίως σημεία που έχουν απομείνει από την Τόχα στον Buenos Aires που προσπαθήσαμε να έχουμε μια νέα συμφωνία, αποτύχαμε. Και καθότι είναι δύσκολο να έχουμε πολυμερή αποτελέσματα, η νέα λεωφόρος για να προχωρούμε είναι plurilaterals. Επί τη βάση των MFM. αυτά που συζητούμε με τους Αμερικανούς και τους Ιάπωνες στα, στα τριμερή για παράδειγμα που τελικώς θα πρέπει να παράσχουν την, ε, το θεμέλιο για την επανεξέταση των κανόνων ή για νέους κανόνες των ΠΟΕ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μία ε, προσέγγιση plurilateral Εν πάση αυτή θα είναι μια υποψήφια τριμερής για την προσέγγιση του plurilateral. Τώρα για την ε, ανάπτυξη του δυναμικού έχετε δίκιο με αυτά που σημειώσατε. Υπάρχει ένα θέμα στον ΠΟΕ εδώ για την βελτίωση την ανάπτυξη του δυναμικού και για το, για το δυναμικό που έχουν τα μέλη να συμμετέχουν. Αυτή τη στιγμή στον ΠΟΕ είμαστε σε μια πολύ εντατική περίοδο τα μέλη ε, καλούνται να απαντούν εντός μίας ή δύο εβδομάδων και υπάρχουν πολλές ομάδες χωρών ή χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Αν ζητήσετε από την Αφρικανική Ένωση σχολιάστε την πρότασή μας, αν λάβουμε οποιοδήποτε σχόλιο εντό ε, πέντε μηνών θα είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Πολλές από τις ομάδες αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα στη Γενέβη στις πρωτεύουσες τους να συζητούν τα θέματα αυτά με επιχειρησιακή διάσταση. Και επομένως αυτές τις πολυμερείς ε, συναντήσεις υπάρχει μια τέτοια ευκαιρία. Για τα μέλη τώρα των ε, σωμάτων έφεσης, των δικαστηρίων έφεσης οι Αμερικανοί λένε ότι αυτοί είναι επιλητές διαφορών, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους γρήγορα και το τελευταίο που θέλουμε είναι ακόμα περισσότερη επέκταση των σωμάτων αυτών γιατί τότε θα γίνουν περισσότερο στα δικαστήρια γι' αυτό δεν το θέλουμε λένε οι Αμερικανοί για το έλλειμμα δημοκρατίας έχετε απόλυτο δίκαιο όπου έχει τέτοιο έλλειμμα Εξού και δημιουργήθηκε το δημόσιο φόρουμ και η κοινοβουλευτική συνεισφορά προς τη δουλειά του ΠΟΕ, προς το έργο του ΠΟΕ έχει ακόμα πολύ δρόμο. Μέχρι την επόμενη υπουργική είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε Και παρότι 15 μήνε απέχουμε από τη συνάντηση αυτή, αυτό δεν είναι πολύ χρόνο για τον ΠΟΕ. Ευχαριστώ και τους δύο για αυτή την ε, συνεισφορά σα Ε, είμαστε πεπισμένοι ότι θα συνεχίσουμε πέρα τη συζήτηση από για αυτό το θέμα. Θα σας ξαναδούμε λοιπόν. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Next item is the joint debate on... Το επόμενο θέμα μας είναι η κοινή συζήτηση στα θέματα 4 και 5 που έχουμε. Μία από τις θέσεις είναι να μην αρχίσουμε διάλογο σε επίπεδο Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Και υπάρχουν και οι σχετικοί κανονισμοί. Αυτά όλα που είχαμε κάνει ήταν βασισμένοι στην κοινή θέση των τριών θεσμικών οργάνων για το 2014. Τώρα, το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να έχει ε, μια νέα εντολή για να μπορέσει να διπραγματευτεί. είναι κρίμα και ντροπή. Διότι αυτό χρησιμοποιείται από κάποιες φταρικές κυβερνήσεις ώστε να αποδυναμωθεί η θέση μας. Είναι λοιπόν απίστευτο το ότι δεν μπορεί να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι σε θέση το Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την ε, σχετική εντολή. Και εγώ και ο πρέσβης στείλαμε μία επιστολή σε όλους τους πρέσβεις ώστε να μπορέσει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, διότι μας απασχολεί αυτή η κατάσταση. Δεύτερον, ζητάει η Επιτροπή να υπάρχει σαφής διαδικασία για την ε, εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, ώστε να υπάρχει ένας κατάλογος με απόλυτη σαφήνεια. Αυτό είναι θέμα ε, πήγων. Υπάρχει ενδιαφέρον από το Συμβούλιο και θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα και θα πρέπει να, τε, να μπορέσει το πακέτο αυτό με τις διάφορες προτάσεις που περιλαμβάνει να ε, επικαιροποιηθεί. Ο κύριος Μπούχνερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Τέσσερα λεπτά άλλωστε έχουμε μόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πω ότι εσείς αναφερθήκατε στα βασικά θέματα. Θα ήθελα όμως και εγώ να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Έχουμε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε και μάλλον δεν θα είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια αυτής της ηττίας να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Αυτό εις βάρος των κοινών μας αξιών. Ήδη αναφέρατε ότι χρειάζεται επιγόντως να κάνουμε κάτι, διότι καθημερινά συλλαμβάνονται άνθρωποι με ευρωπαϊκή τεχνολογία στα χέρια τους. Κάθε μέρα που καθυστερούμε, στοιχίζει την ελευθερία, αν όχι τη ζωή, σε κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ρουμανική Προεδρία για τις προσπάθειές της. Διότι θέλησε να πετύχει κάτι, αλλά αντιμετώπισε την γενική αντίθεση του Συμβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτά που είπατε εσείς να προσθέσω την δική μου απογοήτευση. Να προχωρήσω και στο επόμενο. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται εάν ε, έχουμε τελικά ασπυρό Brexit, Brexit χωρίς συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τρίτη χώρα, ως οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα. Δηλαδή και οι εξαγωγές επικοινωνιακού υλικού δεν θα είναι δυνατές. Αυτό ε, διότι αυτές οι τεχνολογίες συνδέονται στενά με τις ε, τεχνολογίες παρακολούθησης. Αυτό δεν θα είναι καλό ούτε για τη δική μας οικονομία, ούτε για το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι πεπισμένος ότι η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ αυστηρό όσον αφορά τους ελέγχους εξαγωγών. Πρόκειται για τη χώρα όπου είχαμε τις περισσότερες ε, απορρίψεις αιτήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι με ήσυχη τη συνείδηση μπορούμε να βάλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην κατηγορία των χωρών προς τις οποίες μπορούμε να εξάγουμε χωρίς ε, σημαντικούς ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο ε, στους και στον Ε, στο όνομα του κ. Φιέλνερ. Ε, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, σκιώδης εισηγητής μας είναι ο κύριος Φιέλνερ και το, Ινωμέ... το ΕΛΚ στηρίζει τον κανονισμό για ε, την γενική άδεια εξαγωγής για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Ε, όσον αφορά τη μη διάδοση όπλων, ε, την ασφάλεια και τα διεθνή πρότυπα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει σημαντικός εταίρος. Επιπλέον, όσον αφορά την κυβερνοπαρακολούθηση, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αξιόπιστη χώρα. Κατά την αναδιατύπωση του κανονισμού για τη διπλή χρήση θα θέλαμε να πούμε το εξή. Ε, το και μένει στον συμβασμό που επιτεύχθη στο Κοινοβούλιο και που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια πολλά θέματα, όπως ο αυτόνομος κατάλογος, η ρήτρα catch-all και η εξοεδαφική προσέγγιση. Είναι θέματα που δεν μας αρέσουν ιδιαίτερα. Γνωρίζουμε όμως ότι επρόκειτο για συμβιβασμό με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Λυπούμαστε που το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να συμφωνήσει πάνω σε εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε διότι είχαμε διαπραγματεύσεις σε ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη. Οι μακροσκελείς διαπραγματεύσεις έχουν εμποδίσει ε, την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πραγματικής προόδου. Εάν ε, είχε συζητηθεί στην ε, ομάδα εργασίας εξωτερικού εμπορίου το θέμα αυτό που ε, συναντιέται πιο συχνά. θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Ωστόσο, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβληματιστεί. Συμφωνούμε ότι αποτελεί πρόβλημα το να, καταλήξουν, ε, να καταλήξει υλικό κύβερνο παρακολούθηση σε λάθος χέρια. Μήπως ε, θα ήταν καλύτερο να έχουμε ξεχωριστό κανονισμό για τον ε, έλεγχο εξαγωγών αυτών των προϊόντων. Άλλωστε, ο βασικός λόγος ε, των ελέγχων εξαγωγής είναι η μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, κάτι που δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το υλικό παρακολούθησης. Μάλιστα είναι δύσκολο να συγχωνεύσουμε αυτά τα δύο είδη ε, ελέγχων εξαγωγής. Ε, θα πρέπει να ε, εκπονήσουμε την πρόταση για την εξαγωγή αυτών των προϊόντων. Θα πρέπει όμως να έχουμε και μια σωστή πρόταση και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για να έχουμε ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από τους πράσινους η Χάιντι Χάουταλα. Πρόεδρε, απλώ θέλω να πω ότι την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια ζητήθηκε το θέμα αυτό από την Φινλανδική Προεδρία που είναι η επόμενη και μέρος της Τρόικα. Αν κάνει κάτι για την πρώτη θύση αυτή της ε, νομοθεσίας. Δεν απάντησε την ερώτηση, την συνερώτηση όμως του ε, ε, εισηγητού μας, του είπε ότι δεν είχε σχέση. Ο επόμενος ομιλητής, την ΚΟΕ, χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Σας ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους της CR. Εκφράζει την λύπη του, διότι δεν μπορεί στο Συμβούλιο να βρει εντολή για να διαπραγματευτεί το θέμα αυτό που αφορά τα είδη διπλής χρήσεως. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η κυβερνοασφάλεια και η κυβερνοεπιτήρηση διότι φοβόμαστε ότι δεν θα είμαστε σε θέση να εξυγχρονίσουμε τα θέματα ελέγχου για αυτού του είδους τα αγαθά. Επίσης, βλέπουμε ότι ο φάκελος αυτός δεν προχωράει, πράγμα το οποίο θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν μπορούμε οι παρούσες διατάξεις να παραταθούν περαιτέρω. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνούμε με το χρονοδιάγραμμα για την ουσία της πρότασης η οποία έχει υποβληθεί για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ ο Χέλμουτ Σόλτ. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Όχι μόνο πρέπει να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας, αλλά να εκφράσουμε με σαφήνεια το ότι δεν δεχόμαστε αυτή την προσέγγιση του Συμβουλίου. Διότι για ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν υπάρχει καμία συνεργασία. Μπλοκάρεται το θέμα. Θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο λοιπόν να είναι πολύ πιο διαφανές σε αυτά που κάνει για να ξέρουμε ποιο είναι αυτός ο οποίος ε, ε, απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία με εμά, ώστε να προσέχουμε να προχωρήσουμε. Ελπίζω ότι η Ρουμανική και μετά η Φινλανδική Προεδρία θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ολοκληρωθεί τώρα θέμα. Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, όντω πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα υπάρχει το Brexit, αλλά τελικά νομίζω ότι θα πρέπει με σαφήνεια να ορίσουμε τα θέματα τα οποία μας απασχολούν τώρα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία λύση και μία σαφή εικόνα. Και ποιες είναι οι δυνατότητες που θα έχουμε ώστε να είναι ομαλές και στο μέλλον το Ηνωμένο Βασίλειο με μας. Ελπίζω ότι θα συνεισφέρει στου δύο περίπου επόμενους μήνες το Ηνωμένο Βασίλειο για να βρεθεί λύση. Από την Επιτροπή η κυρία Σαμπάρτα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίδετε το λόγο για το θέμα αυτό. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία, βεβαίως η Επιτροπή εκφράζει την λύπη τη διότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να προχωρήσει και να ολοκληρώσει η θέση. Άρα νομίζω ότι στην παρούσα θητεία δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το όλο θέμα αυτό. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Βεβαίως είναι το πουλ απόλυτα πόσο σημαντικό είναι ο φάκελος αυτός. Και σε σχέση για την προώθηση των αξιών του Ευρωπαϊκή Ένωσης, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ε, πολιτικές αλλαγές για τις εξαγωγές, δεδομένου του κακού κλίματος μεταξύ Πακίνας. Τώρα, νομίζω ότι θα μπορέσει τελικά να καταλήξει σε θέση το Συμβούλιο. Δεν είναι τόσο επί της οι διαφορές, αλλά όσον αφορά τη διαδικασία. Και ελπίζω ότι με τη βοήθεια της Ρουμανικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές και τις συμφωνίες που υπάρχουν τώρα για τη δεύτερη νομοθετική πρόταση που αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε γνώμονες και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που προχώρησαν ταχύτερα αυτή την διαδικασία. Ξέρουμε ότι υπήρχε επίγον χαρακτήρας και αυτό είναι κάτι που αναγνωρίστηκε ευθύ εξ αρχής και σας ευχαριστούμε διότι με τη συνεισφορά σας θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα σε αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν είναι κανείς εκ μέρους Συμβουλίου εδώ και αν θέλει να μας εξηγήσει γιατί δεν είναι σε θέση να αναλάβει αυτή την εντολή. Κρίμα και ντροπή, λέει ο πρόεδρος. Και δεν θέλω να ακούσω τίποτε για εμπόριο που βασίζεται σε αξίες και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ντροπή, μην μου ξανάρθει με τέτοια επιχειρήματο το Συμβούλιο. Τώρα, υπάρχουν τροπολογίες. Δεν υπάρχουν τροπολογίες για να μπορέσει ε, να τεθεί στις ε, ασφαλείς χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να το προχωρήσουμε αυτό σύμφωνα με το άρθρο 50 του καταστατικού. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Άρα φτάνουμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Indeed, point six, the... Στο σημείο 6 λοιπόν. Η αλλαγή εξοδότηση, τροποποίηση εξοδότησης για, τα, για ορισμένα είδη διπλή χρήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουμε μια δοκιμή όμως, σας παρακαλώ, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote closed. Πέρασε. Εντάξει, όλα καλά τα βλέπω. Καλά δουλεύει το σύστημα. Έχουμε μία και μόνη ψήφο. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. And the vote is closed. Πέρασε. Ομοφόνος. Στο 7. Η σύναψη των ε, συμφωνιών υπό το άρθρο 11 της GATS και εδώ μία και μόνη ψήφος ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε. And Με μία αποχή. Εγκρίνεται. Στο 8. Το πρωτόκολλο που αφορά στην προσχώρηση της Κροατίας άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ και εδώ μία ψήφος. And the vote is Πέρας, επίσης με ευρύτατη πλειοψηφία, στο 9, το νέο, η, νέα συμφωνία πλαίσιο με την Ελβετία, όπου έχουμε κάποιες δομπολογίες, η συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1α υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική όχι. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 23 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 26 και 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 και 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε το 38 παρακαλώ. Πέρας. Πράγματι απορρίπτεται. Και τώρα ψήφος για το σύνολο της σύστασης. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ όλους. Αυτή ήταν και η λήξη της ψηφοφορίας και πάμε στο σημείο 10. Εάν κάποιος θέλει να αποχωρήσει, παρακαλώ να το κάνει σιωπηρά και ήσυχα. Το σημείο 10 αφορά τις συστάσεις για την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ε, δώσω την Προεδρία, διότι εγώ είμαι μόνιμος συζητητής ε, για εμπορικά θέματα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ξέρετε, πριν δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σχέδιο δύο εντολών διαπραγματεύσεων για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβάζοντας ε, τις εντολές αυτές, δεν μπορούσα να καταλάβω ποια στρατηγική κρύβεται πίσω από αυτές. Από τη μία φαντάζομαι ότι η στρατηγική θα μπορούσε να είναι να ε, αποφύγουμε την κλιμάκωση και ε, να αποφύγουμε εμπορικές διαμάχες. Από την άλλη όμως, υπάρχουν και κάποια στοιχεία στις εντολές αυτές, που νομίζω δεν είναι πολύ σαφή. Να αναφέρω κάποια από αυτά. Καταρχάς, ε, πάντα στο παρελθόν λέγαμε και το έχει γράψει επανειλημμένα ο τύπος αυτό, ότι δεν θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις υποπίεση. Έχουμε ακόμα τα τέλη, τους δασμούς για το ατσάλι, για το αλουμίνιο και έχουμε επίσης και την απειλή δασμών ε, για αυτοκίνητα και ανταλλακτικά. Υπάρχει ο εμπορικός νόμος 232 και δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορία. Από την άλλη, από τις ΗΠΑ δεν έχουμε καμία δέσμευση να ε, εξαλείψει την απειλή αυτή, να άρει ε, τις απειλές αυτές. Έχουμε λοιπόν την αρχή να μην ξεκινάμε ε, διαπραγματεύσεις υπό απειλή, υπό, ναι, και τώρα λέμε ότι θα τις ολοκληρώσουμε, δηλαδή σαν να έχουμε αλλάξει στάση. Δεύτερον, δεν έχω καταλάβει πολύ καλά η εντολή αυτή καλύπτει και τα οχήματα και τα ανταλλακτικά ή όχι. Στην εντολή λέει ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Γιούνκερ της 21ης Ιουλίου. Στην συμφωνία αυτή αποκλείονται ρητά τα οχήματα και τα ανταλλακτικά. Ο Ζωάλη ανέφερε εδώ στην Επιτροπή μας ότι δεν είναι πολύ σαφές αυτό ή ίσως να συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τώρα ποια είναι η επίσημη θέση. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. διότι τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αντιπροσωπεύουν το 1 τρίτο των βιομηχανικών προϊόντων. Εάν αφαιρέσουμε τα αυτοκίνητα από τις διαπραγματευτικές εντολές αυτές, αυτό σημαίνει πρώτον ότι τα βασικά κέρδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συμπερίληψη ε, των αυτοκινήτων ε, δεν ε, θα υπάρχουν πια και πιθανότατα να έχουμε απώλειες και σε άλλα βιομηχανικά είδη. Αυτό βασίζεται σε μελέτη αντικτύπου στο πλαίσιο της διαδικασίας TTIP. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μελέτη αντικτύπου για τούτη την την πρόταση. Μάλιστα υπάρχει νέα προσπάθεια ε, διερευνητικής μελέτης, ε, το scoping exercise. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος αν εξαιρεθούν τα αυτοκίνητα, αυτό να ωφελήσει αποκλειστικά την αμερικάνικη πλευρά. Και δεύτερον, εάν αποκλείονται τα αυτοκίνητα, τότε ο όγκος των δασμών θα βρίσκεται κάτω από το 90%, κάτι που αποτελεί την προϋπόθεση για να έχουμε εμπορική συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΓΑΤ, Η Κομισιόν πάντα λέει ότι το άρθρο 24 απαιτεί τουλάχιστον το 90%. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα συμμορφούμαστε λοιπόν με τον ΠΟΕ εάν δεν φτάσουμε το 90%. Τρίτον, αγαπητοί συνάδελφοι, πάντα λέμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τους δασμούς, αλλά και τους κανόνες που είναι σημαντικοί για το δίκαιο εμπόριο. Το θέμα της βιωσιμότητας δηλαδή μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως και το θέμα της ε, περιβαλλοντικής συμφωνίας του Παρισιού, της συμφωνίας για το κλίμα. Πάντα λοιπόν λέγαμε ότι θέλουμε να γίνεται αναφορά της συμφωνίας του Παρισιού και θέλουμε και σωστή εφαρμογή στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας. Αυτό εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο. Με μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία και με πολύ σαφή διατύπωση στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Έχουμε λοιπόν κάποια σημεία αναφοράς, έχουμε το ψήφισμα TTIP, έχουμε το ψήφισμα του περσινού Ιουλίου έχουμε και κάποιες άλλες σαφείς δηλώσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με το πώς θα πρέπει να διατυπώνονται οι εμπορικές συμφωνίες. Ακριβώς για αυτό το λόγο αμφιβάλλω ότι οι προτινόμενες εντολές πληρούν ε, τις προϋποθέσεις ε, του Κοινοβουλίου. Δίνω λοιπόν τώρα το λόγο στους κοιόδες συζητητές. Χώτε Λίφε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και και σας ευχαριστώ και ως εισηγητή. Είναι λίγο κρίμα, μάλλον είναι πολύ κρίμα το ότι πρέπει να εργαστούμε έτσι υποπίεση. Θα πρέπει ήρεμα να κάτσουμε και να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό πιο χαλαρό κλίμα, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρωπαϊκή πλευρά. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεύτερη παρατήρηση. Αυτά που αναφέρονται εδώ και αυτά που είπατε κι εσείς είναι όλα εκτιμήσεις. Ποιος αποφασίζει. Άλλωστε μπορεί κανείς να δει και με άλλα πολιτικά γυαλιά το κείμενο αυτό. Άλλωστε, ε, δεν είναι κρυφό ότι εμείς ως ΕΛΚ βλέπουμε διαφορετικά κάποια θέματα. Καταρχάς δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε τους κινδύνους εκεί όπου δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ε, αρκετά σημεία στα οποία συμφωνούμε. Επί της αρχής, ωστόσο, το ΕΛΚ πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να κλείσουμε την πόρτα. θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ξέρω τι κείμενα έχουμε εγκρίνει. Θέλουμε να επανέλθουμε σε όσα εγκρίναμε στο τέλος της προηγούμενης θητείας. Αυτό δεν έχει νόημα, διότι η κατάσταση αλλάζει συνεχώς. Δεν βρισκόμαστε πια στον περσινό Ιούλιο. τότε λάβαμε σαφή απόφαση, βρισκόμασταν όμως σε διαφορετική θέση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε διαφορετικά τα πράγματα τώρα. Καθημερινά αλλάζει ο κόσμος, θα πρέπει να προσέξουμε να μην κοίταμε τόσο πολύ τον εαυτό μας που να μην μπορούμε να ακολουθήσουμε. Τι φαντάζεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς βλέπουμε την πρόταση. Νομίζω ότι με κάποιες τροπολογίες και με μια κριτική ματιά θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κλείσουμε την πόρτα και να φροντίσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να Έχουμε διάλογο με τους Αμερικανούς. Και μάλιστα να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στους τομείς όπου συμφωνούμε. Ναι, τα πράγματα δεν είναι τέλεια, σύμφωνα και εγώ, αλλά νομίζω ότι ως κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σαφή θέση και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε κατόπιν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ECR. So, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φανταστείτε... Miss McClarkin, because I will speak on behalf... Φανταστείτε με κυρία Μακλάκλιν, θα μιλήσω εκ μέρους της. Δεν είναι εύκολο να το φανταστείτε αυτό βέβαια, το ξέρω. Λέγει η κυρία Μακλάκιν. Πάντα ήμουνα υπέρ της εμβάνθησης των ε, ε, κανονισμών και των σχέσεων που αφορούν τις ατλαντικές μας σχέσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαιτίας των ε, δις που αφορούν τις συναλλαγές στο εμπόριο και τις εξαγωγές μεταξύ ημών και ημών είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μας βρίσκονται σε δυσκολία. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ε, διαπραγματευόμαστε υπό διακατεχόμενοι από το αίσθημα του φόβου. Πρέπει όμως να δούμε κατά πόσον θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτά τα οποία συνεφώνησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο ε, Γιούνκερ. Πιστεύω ότι θα πρέπει λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν για τους δασμούς που αφορούν καταρχάς τον ε, σίδηρο και, τον, ε, και το ατσάλι, αλλά δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε περαιτέρω υποχωρήσεις για δασμούς σε άλλα προϊόντα. Ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ ψηλούς δασμούς ε, η Αμερική για κατεργασμένα προϊόντα. Σε αυτούς τους τομείς ε, η κατάρριξη των δασμών θα ανοίξει νέους δρόμους για τους εξαγωγείς μας και θα μπορέσει να αυξήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας και οι μιμία μας θα υποφεληθούν από την ε, όλα αυτά τα, την χαρτούρα προσυρμόρφωση, τα πιστοποιητικά και όλα τα εμπόδια. Πιστεύω ότι δίδεται μία, γίνεται μία σαστή απεικόνηση ως στον παρόντο κανονισμό όλων των στοιχείων που αφορούν την περούσα κατάσταση και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένες αποφάσεις από αυτού του θέματος. Πιστεύουμε ότι όμως θα πρέπει να δούμε την κατάσταση ε, και δεδομένη της παρούσας κατάστασης διεθνώς να ξαναρχίσουμε διαπραγματεύσει ώστε να αποκλιμακωθεί το ψυχρό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί για να βοηθηθούν όλες οι βιομηχανίες και ημών και ημών. Ελπίζω ότι με το ψήφισμα αυτό θα επιτραπεί στις ε, βιομηχανίες να να μπορέσουν σε θέματα συμμόρφωσης, πιστοποίησης και ό,τι αφορά τις μικροσωματικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν, θα πρέπει το θέμα αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσουμε όλοι με μία ενιαία φωνή για να προσχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ και να βρούμε την μέση οδό, την οδό της ναι. λογικής για να προχωρήσουμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό περαιτέρω και με τον εισηγητή και τους ε, άλλους συνηγητές ε, για, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Σόλτς για, ε, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα συμφωνήσω με, την, με τα πολύ προσεκτικά σας σχόλια σχετικά με την εντολή αυτή. Μέσω της επιταχυμένης διαδικασίας ε, στο Κογκρέσο, τα πράγματα έχουν πιεστεί. Και η επιταχυμένη αυτή διαδικασία κατευθύνεται προς το, ε, την μελλοντική σχέση ε, με τους Αμερικανούς ε, και αναφερόμαστε στα γεωργικά προϊόντα τελεία. Τόσο ξεκάθαρα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς η Κομισιόν, από πού βρήκε την ιδέα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αυτές υπό το πλαίσιο αυτό. Έχουμε αλουμίνιο, χαλιβουργία, βρισκόμαστε στην ίδια στο ίδιο τέλμα που βρισκόμασταν ε, ε, εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή θεωρούμε μήπως ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης οι κόκκινες γραμμές θα αρθούν. Γιατί κανείς δεν ξέρει αν ο Τραμπ θα σεβαστεί αυτές τις κόκκινες γραμμές θα βρεθούμε μήπω να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση αντίστοιχη με τη TTIP ή μήπως ε, πρέπει να σκεφτούμε, να αναλογιστούμε ποιος είναι ο στόχος τελικός αυτής της εντολής, σε τι θα χρησιμοποιηθεί. Τα δασμολογικά 3 σε 4% δεν είναι τόσο το πρόβλημα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που τι ενδιαφέρει τι επιχειρήσει είναι η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά των κρατών μελών. Και γνωρίζουμε την ομοθεσία Οι αμερικανικές επιχειρήσεις όμως θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στην ε, ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Έτσι, οι συνθήκες ανταγωνισμού διακυβεύονται και έτσι και οι θέσεις απασχόλησης. Συμφωνώ δηλαδή μαζί σας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν την βιομηχανία, τα προϊόντα. Δεν μπορούμε απλά να πούμε ότι ωραία θα καταργήσουμε τους δασμούς. Πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην κοινωνία, στην απασχόληση, στην καθημερινή ζωή. Και επίσης ε, από την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λείπει τελείως ένα κεφάλαιο βιωσιμότητας. Θυμάμαι ότι ήταν επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υπάρχει τέτοιο κεφάλαιο σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες. Και τέλος... Είναι πολύ σημαντικές οι διακλαντικές σχέσεις, το γνωρίζουμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, έχουμε τη θέση του Κοινοβουλίου, πρέπει όμως να έχουμε αξιοπιστία στην όλη διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν τα Εθνικά Κοινοβούλια να συνομιλήσουν με τους υπουργούς τους και έτσι θα μπορέσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να εργαστούμε επικοδομητικά. Έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο και συμφωνώ με την Κότελίδε. Βεβαίω και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο συζητείται και σε επίπεδο εθνικών ε, κοινοβουλίων. Η Μαρία Ρένα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε ως εισηγητής για την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε. Δηλαδή, είπα και Ιδιαίτερο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν σέβονται το ε, νομικό πλαίσιο του ΠΟΕ. Και είναι παράνομοι οι δασμοί τους οποίους ε, προβάλλουν. Δεν σέβονται ούτε την πολυμέρεια, ούτε τους διεθνείς κανόνες και ξέρουμε ποια είναι οι ιδέες του Τραμπ ή σε επίπεδο ΠΟΕ είτε σε επίπεδο συμφωνίας όσον αφορά την COP21 και 24 όσον αφορά το κλίμα. Επίσης, διαρωτώμε πώς θα μπορούσαμε να συμβιλιώσουμε την προσφορά που γίνεται σήμερα στα πλαίσια της εντολής του σε Επιτροπή για το Συμβούλιο και την προσφορά της Αμερικανική κυβέρνηση. Βλέπω ότι υπάρχουν απολύτω διεστάμενε απόψεις μεταξύ αυτών των δύο προσφορών. Αν υπήρχαν κάποια κατελάχιστον κοινά σημεία θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε συζήτηση. Δεν υπάρχει όμως τίποτε αν δούμε τι προσφέρει ο καθένα και κυρίως είπα. Διερωτώ με λοιπόν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα σήμερα να ε, υιοθετήσουν αυτή τη ε, διαδικασία fast track και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Δεν έχει γίνει καμία σχετική μελέτη επί του θέματος. Επίσης, σε μία τοποθέτηση στην οποία θα πρέπει να ισχύουν τρεις προϋποθέσεις πριν να προχωρήσουμε. Τι ισχύει. Πρώτα απ' όλα, οι δασμοί που προτείνει η, η που δεν έχουν καμία σχέση με τους κανόνες του ΠΟΕ θα πρέπει να αρθούν. Δεύτερον, Δεύτερη προϋπόθεση, απαραίτητη. Θα πρέπει είπα να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις που αφορούν το κλίμα. COP21 και 24, δεδομένου ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κυρώσεις για τις επιχειρήσεις μας, που λαμβάνουν μέτρα και, και τα μέτρα αυτά έχουν αντίκτυπο για αυτές. Και απ' την άλλη έχουν ανταγωνιστεί κάποιον ο οποίος δεν δίνει δεκάρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Άρα εδώ υπάρχει αντίκτυπος αρνητικός θα δημιουργήσουμε δυσκολίες για τις επιχειρήσεις μας στην Ευρώπη. Το ΕΛΚ και το ECR που πρέπει καταρχήν να προασπίζονται τις επιχειρήσεις, τις αφήνουν χωρίς καμία προστασία μπροστά στους ανταγωνιστές. Διερωτώ με, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που θα βάλουν κάποια στιγμή και το ECR και το ELK σε θέματα εμπορικά. Θα πούν κάποια μέρα ότι αρνούμαστε να κάνουμε διαπραγματεύσεις. αχύψη ο μεγαλόγους, γιατί αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση του Τραμπ είναι στα άκρα του μη σεβασμού των κανόνων ελεύθερη ανταγωνισμού. Και λένε κάποιοι, παρόλα αυτά θα θέσουμε τις επιχειρήσεις μας σε κατάσταση ανταγωνιστικότητας παρά το γεγονό που είναι άδικο αυτό σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, κυρίως αυτούς οι οποίοι υποκινούνται από τον Τραμπ και δεν σέβονται τίποτε. Όπου και αν βρίσκεται λοιπόν κανείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάποιους κανόνες θα πρέπει να τους σέβεται απόλυτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα για το θέμα αυτό να πω τα εξής. Σωστά. Μια νέα διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ είναι εντελώς αντίθετη με αυτά το οποίο είπε η κυρία Μάλστρομ. Δεν διαπραγματευόμαστε, είπε, αν κάποιος μας βάλει το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν έγινε επίσης καμία μελέτη αντικτύπου. Είναι απαραίτητο αυτό. Ελπίζω ότι αυτό θα συμπεριληφθεί στο ψήφισμα του εισηγητού μας. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε την επιθυμία ε, των ε, ΙΠΑ να πολλούν τα προϊόντα τους επιβάλλοντας δασμούς. Όσον αφορά το TTIP, υπάρχουν μεγάλες ε, ε, ομοιότητες, αλλά μεγάλες διαφορές και με το τι ακριβώς ε, απαιτεί για την ποιότητα των προϊόντων από τους παραγωγούς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ, ε, βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων. Όσον αφορά κάποια άλλα προϊόντα, ε, το εισαγωγή προϊόντων ε, μεταποιημένων. δεν υπάρχει καμία προστασία. Όσον αφορά επίσης την πιστοποίηση συμμόρφωσης, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ε, μια διαδικασία που βασίζεται σε κανόνες, αλλά κάτι που θέλει να εφαρμόσει με ενιαίο τρόπο. Άρα αυτό είναι κάτι που ασκεί πίεση στις δικούς μας κανόνες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά να έχουμε και απαιτήσει ώστε να γίνουν σεβαστά κάποια προϊόντα. Η Κάρολιν, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά την Κομισιόν που έλεγε ότι θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις υποπίεση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνουμε αξιόπιστοι. Οι πολίτες το περιμένουν αυτό από μας. Περιμένουν και ασφάλεια, περιμένουν και εγγύηση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες. Ξέρω ότι θα ήταν λάθος να κλείσουμε την πόρτα απέναντι στις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να εγκρίνουμε διαπραγματευτική εντολή. Είναι σαφές ότι μόνο προς όφελος της Αμερικής θα είναι. Εμείς θα θέλαμε οι εργαζόμενοι μας να ωφεληθούν από μια τέτοια συμφωνία. Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι αξιόπιστος εταίρος. Είτε μιλάμε για τη Συμφωνία για το Κλίμα, είτε μιλάμε για τον ΠΟΕ, βλέπουμε σημαντικές δυσκολίες και δεν βλέπω να έχει νόημα να εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή διαπραγματευτική εντολή. Και να πιστέψουμε αφελώ ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, ότι θα βελτιωθούν και οι σχέσει μας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσματα. Χρειαζόμαστε καλές και διαφανείς εμπορικές συμφωνίες και η Κομισιόν ακολουθεί λάθος κατεύθυνση. Ελπίζω και το Συμβούλιο να μας ακολουθήσει να μην εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή. Αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια άλλη στιγμή και με διαφορετικό είδος διαλόγου. Διάλογος δεν σημαίνει έγκριση διαπραγματευτικής εντολής, σημαίνει να συνομιλήσουμε σχετικά με τις διαδικασίες. Ευχαριστώ κύριε Σφίγκλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πρόεδρο, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουμε λίγο την οπτική μας και να δούμε έχουμε εμπορικό πόλεμο διεθνώς ή όχι. Γιατί μερικοί μελετητές λένε ότι πράγματι έχουμε απόλυτη αντιπαράθεση, άλλοι λένε ότι έχουμε σημάδια καλής διαπραγματεύσης. Είναι, είναι, είναι σημαντικό να διατηρούμε μια διατλαντική σχέση. Φαντάζομαι ότι όλοι εδώ θα συμφωνούσαμε ότι η διατλαντική σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, θέλουμε λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές. Θέλουμε να δούμε ποιο είναι το συμφέρον των επιχειρήσεών μας και των οικονομιών μας. Αν εξετάσουμε την δυναμική των εμπορικών σχέσεών μας με τις Ηνωμένες και με τις υπόλοιπες χώρες, πέρυσι το 18 ήταν τουιτάρισμα απάντηση. Τουιτάρισμα απάντηση. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω. Και επομένως επειδή το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει και ολοκλήρωσέ τους, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε συμφωνία, ούτε ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις. Σημαίνει ότι είμαστε στο τραπέζι, τουλάχιστον σε τεχνικό επίπεδο, μέσω της διαπραγματεύσης της Κομισιόν τουλάχιστον σε ένα διαφορετικό επίπεδο από αυτό του Twitter. Έτσι. Νομίζω ότι ο ερελισμός επιτάσσει να είμαστε ανοιχτοί στις δυνατότητες που, υπάρχουμε, που υπάρχουν. Το να ανοίξουμε κάτι δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το ολοκληρώσουμε εφόσον δεν, δεν θα είναι προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, των υπαλλήλων τους και των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ διπλά για τη δουλειά σας ε, σχετικά με το θέμα αυτό της εμπορικής μας σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, ε, όπως γνωρίζετε, εγώ υπερασπίζομαι την αρχή των σχέσεων επί τη βάση ενός ισόρροπου και δίκαιου εμπορίου. Είμαι υπέρ και της συνέπειας νομίζω ότι στην πολιτική είναι απολύτως απαραίτητο να αναλαμβάνουμε μια τοποθέτηση την οποία να μπορούμε να υπερασπιστούμε έναντι των πολιτών μας και της κοινή γνώμης με απόλυτη διαφάνεια. Στα πλαίσια λοιπόν της διαπραγμάτευσης αυτής της εμπορικής με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Εγώ ήμουν υπέρ μιας διαπραγμάτευσης της TTIP με τη διακυβέρνηση Ομπάμα με όλες τις δυσκολίες που είχαμε τότε. Αλλά το υπερασπιζόμουν διότι επίσης είμαι υπέρ της διατήρησης της σημαντικής διατλαντικής σχέσης, αλλά όχι σε οποιοδήποτε τίμημα και με οποιαδήποτε διακυβέρνηση. Είναι θεμελιώδες οι αξίες να είναι κοινέ. να συμφωνούμε επ' αυτών. Και αυτό δεν το βλέπω καθόλου στη διακυβέρνηση Τραμπ. Υπάρχει μια απόλυτη αντίδραση στην εμπορική συνολικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλούμε μόνο για συγκεκριμένα βιομηχανικά προϊόντα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισίου. Γιατί αν κάτι επηρεάζει την βιώσιμη ανάπτυξη είναι η βιομηχανική παραγωγή. Και αν η βιομηχανική παραγωγή δεν γίνεται υπό τις αξίες και τις αρχές που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, τότε δεν αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή. Που θυμίζω ότι είναι από τους πρωταρχικούς στόχους που υπερασπίστηκε αυτό εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες του οι πολιτικές ομάδες. Επίσης, για να διαπραγματευτείς με κάποιον πρέπει να του έχεις μια κάποια εμπιστοσύνη. Και διαρωτώ με, ο πρόεδρος Τραμπ καλύπτει τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αισθάνεται ασφαλής και να τον εμπιστεύεται. Γιατί μέχρι στιγμής έτσι όπως έχει συμπεριφερθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν με σημαντική έλλειψη σεβασμού. Διατηρώντας υπόψη λοιπόν όλα αυτά συν την υπεράσπιση, την προάσπιση του, της πολυμέρειας, κάτι που επίσης ενέκρινε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία των, μεταξύ των πολιτικών ομάδων, το εμπόριο δηλαδή, που βασίζονται στις αρχές και τους κανόνες του πολυμερούς εμπορίου και των πολυμερών σχέσεων. Το οποίο επίσης είναι κάτι που ε, ε, δεν προσυπογράφει ο πρόεδρος Τραμπ. Επομένω, υπό τι συνθήκε αυτές, τι είδου ε, ε, διαπραγματευτική εντολή θα ήταν αυτή. Νομίζω ότι θα υπήρχαν πολλοί λόγοι για να μην προχωρήσουμε προς την ε, κατεύθυνση αυτή και συμφωνώ με τη συνάδελφο. Ναι, ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι η εντολή αυτή πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τον κύριο Γιούνκερ ε, που έχει την τάση να διαπραγματεύεται και να συζητάει χωρίς καμία εντολή. Το πλαίσιο αυτό αντίθετα πιστεύω ότι πηγαίνει προς μια σωστή κατεύθυνση με δεδομένε βεβαίω τι ανησυχίε των πολιτών. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει όμω επ' αυτού. Καταρχά, εκπλήσωμαι κάπω ε, από τον άτυπο χαρακτήρα αυτής της ε, Κομισιόν. Αυτό το ψήφισμα που είναι αρκετά επιθετικό προς τη διακυβέρνηση του Τραμπ και που θα μπορούσε να έχει και πολιτικά υπονοούμενα πίσω από αυτό το καλό κείμενο. Επίσης το ψήφισμα αυτό μας βοηθάει να σκεφτόμαστε ότι ίσως δεν είναι υπέρ της προάσπισης των επιχειρήσεων και των πολιτών μας και της οικονομίας μας, αλλά περισσότερο για να θίξει, να ντροπιάσει αυτόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Όλα, όλα τα σχόλια που έχουν γίνει για το άδικο εμπόριο, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κτλ. δεν μας φαίνονται ε, να γίνονται σε, στα πλαίσια άλλων συμφωνιών ελεύθερης, ε, ελευθερών συναλλαγών. Εδώ αρνούμαστε τη διαπραγμάτευση ε, υπό τις επιταγές του ΠΟΕ στα πλαίσια ενός πολυμερούς εμπορίου προς το οποίο δεν συμφωνούμε απολύτως. Τώρα αναφερθήκατε στη στρατηγική. Αλλά τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Μήπως πίσω από αυτή τη στρατηγική ε, κρύβονται έτσι ψηφοθυρικές ε, προσεγγίσεις. Εμείς θα έχουμε υποστήριξη σε αυτήν την πρωτοβουλία, επικριτική, αλλά υποστήριξη. Προσεκτική δηλαδή, αλλά υποστήριξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ούμπεν ε, από, εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα και από πλευράς μου δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις προς εσάς. Τα αυτοκίνητα είναι μέσα στην συμφωνία ή όχι. Γιατί αν είναι μέσα, αν συμπεριλαμβάνονται, τότε η απειλή πρόσθετων δασμών μάλλον μειώνεται. Επίσης, είχα πολλές επαφέ με εκπροσώπους τη της ε, βιομηχανία τι τις τελευταίες και μας είπαν ξεκάθαρα ότι η αυτοκινηστική βιομηχανία πρέπει να συμπεριληφθεί. Διότι αλλιώς το συνολικό αποτέλεσμα θα ήταν πραγματικά ελάχιστο. Το οποίο με οδηγεί στο δεύτερο ερώτημα. Ποιο είναι ο αντίκτυπος, ποιο θα είναι ο αντίκτυπο. Έχετε κάποιε ενδείξει του ποιο θα είναι ο αντίκτυπο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία της εντολής αυτής. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω εισαγωγικά κάποιες παρατηρήσεις για να σας εξηγήσω το πλαίσιο εντός του οποίου υποβάλαμε στο Συμβούλιο την εντολή πριν από δύο εβδομάδες. Μια εντολή την οποία συζητάτε και εσείς τώρα σε προετοιμασία του ψηφίσματός σας. Εξελέγει ο πρόεδρος Τραμπ, ξεκίνησε αυτή την πλατφόρμα οικονομικού εθνικισμού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της Προεδρίας του ακούσαμε τη ρητορική του και τις διάφορες θέσεις του, ενώ πέρσι το 2018 ελήφθησαν τα πρώτα εμπορικά μέτρα, τα οποία ε, είχαν αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό εμπόριο χάλιβα. Αρχίσαμε τη συνομιλία με τους ομολόγους μας ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά παρόλα αυτά επέλεξαν να επιβάλλουν δασμούς σε εξαγωγές ευρωπαϊκές προς τις Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι, έτσι Ιούλιο πέρσι εφαρμόσαμε και εμείς αντισταθμιστικά μέτρα. Μέσα Φεβρουαρίου Λίγη το καθεστώ για τα οχήματα. Θα πρέπει να δούμε τότε τι θα γίνει με τις κατευθυντήρε γραμμές, αν θα δημοσιευτούν. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προθεσμία που απέχει μέρες μόλις. Στο πλαίσιο αυτής της νέας έρευνας είχαμε μακρά συζήτηση στο περιθώριο του G7 στον Καναδά τον Ιούνιο. Οι περισσότεροι από εμά το θυμόμαστε αυτό. Αυτό οδήγησε στον αποδεχτή ο πρόεδρος Γιούγκερ την ε, πρόσκληση να πάει στον Λευκό Οίκο. Προετοιμάσαμε την επίσκεψη αυτή μαζί με την Επίτροπο Μάλμστρομ και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν θετικό για τις διαθλητικές σχέσεις. Η συμφωνία αναγνώριζε το βάθος ε, των, ε, των διατλαντικών οικονομικών ε, σχέσεων καθώς και τις προσπάθειες για να έχουμε θετικό θεματολόγιο και να μην καταλήξουμε σε ένα αρνητικό σπιράλ επιβάλλοντας επιπλέον μέτρα πέρα από τη, το, τους δασμούς στο Χάλιβα. Τον Σεπτέμβριο λοιπόν σε διάφορους τομείς εξετάσαμε τους βιομηχανικούς θασμούς, για παράδειγμα στην ενέργεια, τη σόγια και άλλα προϊόντα αρχές Σεπτεμβρίου, ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου λοιπόν και στις Βρυξέλλες και στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, έχουν εξεταστεί τα θέματα αυτά. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυτές τις δύο εντολές ε, προς το Συμβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι ένα θετικό θεματολόγιο ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι προς όφελος της Ευρώπης. αλλά εφόσον υπάρχουν και κάποιες κάποιοι περιορισμοί. Για παράδειγμα, συμφωνούμε ότι ε, μπορεί να έχουμε συμφωνία μόνο εφόσον αρθούν τα μέτρα για το χάλιβα. Είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε συμφωνία για τους βιομηχανικούς δασμούς μόνο εφόσον δεν επιβληθούν μέτρα στα οχήματα, στα μηχανοκίνητα οχήματα ή στα ανταλλακτικά τους. Και να μην έχουμε μέτρα με βάση ε, την παράγραφο 301 ή τίποτα ανάλογο, δηλαδή να μην έχουμε μονομερή μέτρα από πλευράς των Συνωμένων Πολιτειών. Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν κατά διάρκεια των συζητήσεών τους. Η συμφωνία αυτή όμως δεν προβλέπει, όπως είπε και ο πρόεδρος, διαπραγματεύσεις για τον ε, τομέα της ναυτιλίας ή για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Δεν διαπραγματευόμαστε το μορφότυπο της TTIP, δεν πρόκειται για ολοκληρωμένη πλήρη συμφωνία, ούτε είναι η πιο προηγμένη που ε, έχουμε. Δεν πρόκειται για μια μακρά σειρά κανόνων, αφορά συγκεκριμένους τομείς πάνω στους οποίους συμφώνησαν οι πρόεδροι κατά τη διάρκεια ε, μιας πολιτικής και διπλωματικής συζήτησης, ε, κατά τη διάρκεια δηλαδή της επίσκεψης του Προέδρου μας τον Ιούλιο στη Washington. Δύο-τρει συγκεκριμένε παρατηρήσει, κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο του Ιουλίου αποκλείει τα αυτοκίνητα. Έχετε δίκιο, λοιπόν. Λέμε στους Αμερικανούς ότι θέλουμε να σεβαστούμε το κείμενο του Ιουλίου. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πέρα από τα όρια αυτού του κειμένου, όσον αφορά για παράδειγμα τη συμπερίληψη της γεωργίας. Δεν θέλουμε να συμπεριλάβουμε την γεωργία και η γεωργία αποκλείστηκε. Και αυτό είναι κάτι που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημειώνουμε λοιπόν ότι στο κείμενο αποκλείονται και τα μηχανοκίνητα οχήματα και αυτό πράγματι οδηγεί σε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τη συμβατότητα με τον ΠΟΕ, όπως ε, αναφέρατε κι εσείς. Αλλά τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από την εκτελεστική ομάδα εργασίας ε, και ο πρόεδρος Τραμπ επανειλημμένα έχει τουιτάρει σχετικά με τους άδικους δασμούς στα οχήματα στο εμπόριο Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωση. Νομίζω λοιπόν ότι επιδεικνύουμε συνέπεια όταν λέμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, ότι είμαστε διατεθειμένοι να ε, συμπεριλάβουμε όλον τον βιομηχανικό τομέα, ακόμα και τα οχήματα, εάν αναγνωρίσετε ε, από πού ξεκίνησε η διαμάχη, διότι εσείς ξεκινήσατε τις έρευνες για τα οχήματα. Πρέπει λοιπόν ε, να αναγνωρίσουμε την ε, έναρξη του προβλήματος ε, που ήταν η μελέτη για τα οχήματα του Μαΐου. Ο πρόεδρος Γιούνκερ όμως θέλει επίσης να σεβαστούμε τις παραμέτρους που συμφωνήθηκαν ανάμεσα σε εκείνον και τον πρόεδρο Τραμπ. Δεν ξέρω αν αυτά αρκούν ως απάντηση. Διότι Συνεχίζουμε να λέμε ότι αποκλείονται, εξαιρούνται τα αυτοκίνητα, αλλά θα θέλαμε πολύ να συμπεριληφθούν. Θέλουμε όμως οι Ηνωμένε Πολιτείε να αναγνωρίσουν πού ξεκίνησε η διαμάχη αυτή. Ξεκίνησε από τη διαφορά των δασμών. Συμφωνήθηκε επίσης να μην έχουμε πλήρη μελέτη αντικτύπου ε, τη στιγμή υποβολής ε, της εντολή στο Συμβούλιο, διότι η εκπόνηση μιας μελέτης αντικτύπου απαιτεί πολλούς μήνες. Τα έγγραφα αυτά αφορούν πολλές υπηρεσίες της Κομισιόν και οποιαδήποτε μελέτη αντικτύπου απαιτεί 9 έως 12 μήνες. Στο πλαίσιο λοιπόν της ε, συμφωνίας μεταξύ των δύο Προέδρων και γνωρίζοντας ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες ε, από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, θα είναι μέσα Φεβρουαρίου έτοιμε να διαπραγματευτούν μαζί μα. Υπό το φως των πολλών μελετών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ε, απελευθέρωση των διαφόρων τομέων και το διατλαντικό εμπόριο, αποφασίσαμε να παραβλέψουμε την ανάγκη, για, να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για μελέτη αντικτύπου. Υπάρχουν μελέτες εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου εξετάζουμε τα εσωτερικά μας μοντέλα σχετικά με την ε, προσαρμογή ε, των δασμών σε διάφορα βιομηχανικά προϊόντα και εντός εβδομάδων θα μπορέσουμε να σας διαβάσουμε τα στοιχεία. Δεν έχουμε λοιπόν επίσημη μελέτη αντικτύπου. Ε, Έχουμε όμως εσωτερικές ε, μελέτες και είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Πιστεύουμε πάντως ότι οι δύο αυτές διαπραγματευτικές εντολές συνάδουν με το συμφέρον ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, αναζητήσουμε θετικό θεματολόγιο στον τομέα του εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ίσως αυτό οδηγήσει και διαφορετική αξιολόγηση. Αλλά... Αυτό είναι κάτι που θα γίνει στη συζήτηση που θα κάνουμε για το σχετικό ψήφισμα. Σα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ελπίζω ότι θα υπάρχουν τροπολογίες. Η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 6 Φεβρουαρίου. Δεδομένου ότι έχουμε λίγο χρόνο, το ξέρουμε, 6 Φεβρουαρίου. Επίσης, σας υπενθυμίζω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν ότι επιδεδομένου ότι έχουμε έλλειψη χρόνου, όλα θα συζητηθούν μόνο στα αγγλικά. Μόνο στα αγγλικά και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό έδαφος, έδαφος συμφωνίας. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση του σημείου 10 και περνούμε αμέσως στην κοινή συζήτηση των σημείων 11 και 12. Πρόκειται κατά εξοδότηση κανονισμό τη Επιτροπή για τη Συμπλήρωση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μοθολογία και τα κριτήρια εξελόγηση και αναγνώριση συστημάτων δέου επιμέλεια στην αλυσίδα φοδιασμού όσον αφορά κασίτερο, ταντάλιο, βολφράμιο και χρυσό. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει και στην Επιτροπή να συζητηθεί το θέμα αυτό που αφορά την σχετική νομοθεσία που αφορά τα ορυκτά αυτά τέσσερα προϊόντα. Πρόκειται για κανονισμό που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2021. Πάρα πολλά θέματα ακόμη θα πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν πριν από την ημερομηνία αυτή. Οι αρμόδιες αρχές, ε, ε, οι διαδικασίες παραβίασης, ε, κάποια άλλα θέματα που αφορούν ανώτατα, κατώτερα όρια που δεν υπάρχουν ακόμη στον κανονισμό κτλ. κτλ. Προς το παρόν θα ασχοληθούμε με την κατεξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, τον οποίο ελέγχουμε και εξετάζουμε εδώ και την μεθοδολογία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση και των εφοδιαστικών αλυσίδων για τους εισαγωγείς της ε, Ένωσης. Ο κύριος Βίνκλερ, εισηγητής, έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της νομοθεσίας εδώ, στα πλαίσια της θητείας μας. Το Μάιο 17 υιοθετήθηκε ο κανονισμός τα ορυκτά από ζώνες συγκρούσεων. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική να δοθεί η δέουσα επιμέλεια, κυρίως για τους εισαγωγείς μας, για τα τέσσερα αυτά προαναφερόμενα ε, μέταλλα, είχαμε πίεση χρόνου. Η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και οι διάφορες εταιρείες του κλάδου προετοιμάζονται και, προτείνουν και, πρέπει να προτείνουν και διάφορα συνεδευτικά ε, μέτρα στον κανονισμό. Έχουμε συμφωνήσει για κάποια μέτρα, πρόκειται για κανονισμό κατά εξουσιοδότηση και σήμερα κάνουμε τη κοινή συζήτηση αυτών των δύο θεμάτων, διότι πιστεύουμε ότι ο οργανισμός αυτός ο κατενεξιοδότηση, ο σχετικός, θα πρέπει να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και να συζητηθεί στα συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν την προετοιμασία και των κυβερνήσεων και των ε, βιομηχανίας του κλάδου, δεδομένου ότι όλοι έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε σχέση με το θέμα αυτό, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εφαρμοστεί σωστά αυτός ο κανονισμός. Η Επιτροπή μας έχει στείλει τον σχετικό κανονισμό έχει ε, συμπεριλάβει και διάφορους ορισμούς όσον αφορά τις ζώνες συγκρούσεων και τις εμπόλεμες ζώνες, από τις οποίες προέρχονται κάποια προϊόντα. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά από όσον ξέρω μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ ενεργά στο θέμα αυτό θέλουν να προχωρήσουν στην ε, ορισμό της κάθε εθνικής ρυθμιστικής αρχής και η ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων ε, συναντάται σε τακτά διαστήματα για να συζητήσει διάφορα θέματα και το θέμα της εφαρμογής σε κάθε χώρα αυτού του κανονισμού. Επίσης, χαιρετίζω το γεγονός ότι η Κομισιό έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις πολιτικές ή τεχνικές, φέρει πίν, ε, τη μετάφραση των ε, διαφόρων εγγράφων τα οποία ισχύουν σε αφορά τον κανονισμό και σε επίπεδο ΩΣΑ, άλλες τεχνικά θέματα και ελπίζουμε ότι θα είναι προορατική η σχέση που θα υπάρχει ως αναφορά την ε, εποπτεία της εξέλιξης του θέματος αυτός. Σταματώ τώρα και θα ήθελα να δω πώς θα έχει ο διάλογος και με τους ε, συναδέλφους και με την Κομισιό. Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει πώς έχουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Το λόγο τον ε, δίδω τώρα στον κύριο Φρανσίσκο Πέρες Κανάδο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ήταν οπωσδήποτε και χάρη στην ηγεσία αυτού εδώ του σώματος που τον, τον Μάιο του 2017 εγκρίναμε σημαντικό νομοθέτημα που υποστηρίζει την ενωσιακή ηγεσία ιδιαίτερα σε αυτά τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες όπου εδώ προσπαθούμε να, να διαρρήξουμε τη σχέση μεταξύ παράνομων δραστηριοτήτων εξόριξης και της προσπάθειας σταθεροποίησης ε, των συγκρούσεων αυτών και τώρα προσπαθούμε αυτή την προσέγγιση να την ε, κάνουμε πραγματικότητα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις, τις υποσχέσεις που έχουμε αναλάβει εναντί πολλών εταίρων στον κόσμο. Και θα ήθελα να διαβάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η 1η Ιανουαρίου του 2021 μπορεί να φαίνεται πολύ μακριά, αλλά όπως λέμε στα ισπανικά, στην πραγματικότητα είναι μανιάνα, αύριο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι μέχρι την ημερομηνία εκείνη θα έχουμε υλοποιήσει πλήρω τον σημαντικό αυτόν κανονισμό και να δείξουμε με το παράδειγμα, να δώσουμε το παράδειγμα μάλλον με τις πρωτοβουλίες μας, με δύο συγκεκριμένες ρητές δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό, αλλά και συνοδευτικά μέτρα, προς τα οποία είχαμε συμφωνήσει σε πολιτικό επίπεδο, και τα οποία εν πωλής ανταποκρίνονται στις ε, επιταγές του Κοινοβουλίου. Προτού πάω σε λεπτομέρειες για την τον κανονισμό, να πω ότι όπως λέμε και στον κανονισμό των ορυκτών ε, πόλεμων ζωνών, χρειάζονται κατευθύνες γραμμές για τις επιχειρήσεις, ώστε να ταυτοποιούν τις πιο επικίνδυνες περιοχές, ζώνες, και σημαντικές κατευθύνσεις για τους συναδέλφους που θα επιβλέψουν όλα αυτά και θα εξασφαλίσουν ότι όλα αυτά θα εφαρμόζονται σωστά. Χρειάζεται λοιπόν επαρκής και εξαγωγική έλεγχη. Όλα αυτά συνοδεύτηκαν από την επιλογή, τη διαδικασία επιλογής της ε, εξωτερικής ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης που θα μας παράσχει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο των πιο επικίνδυνων εμπολέμων ζωνών στους ερχόμενους μήνες, ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο για να συμμορφωθούμε προς τις διατάξεις του κανονισμού. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα που είναι ο κατεξιότητας κανονισμός και η μεθοδολογία την οποία θα εφαρμόσουμε για τα προγράμματα δέουσας επιμέλειας γιατί αυτό είναι η αρχή ε, για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν. Θα έχουμε και την επίσημη επικύρωση και αναγνώριση των ε, προγραμμάτων αυτών δέουσας επιμέλειας που είναι πολύ σημαντικά για τους εξαγωγείς μας και μετά από αυτό σε μια τρίτη φάση θα έχουμε έναν κατάλογο υπεύθυνων και αξιόπιστων ε, κέντρων επεξεργασίας διεθνώς των ορίτων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν οι συνομοθέτες να έχουν καλυφθεί να είναι ικανοποιημένοι από όλες τι διατάξει αυτέ γιατί αλλιώς δεν θα καταφέρουμε εγκαίρω να υλοποιήσουμε τον κανονισμό. Για τα συνολικά μέτρα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ όχι μόνο στην πρώτη δέσμη μέτρων για, για την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά ιδιαίτερα για τις πολιτικές ε, των της προμήθειας των κατάντι επιχειρήσεων ή στο πεδίο των ρηκτών αυτών. Την άνοιξη φέτος θα δημοσιεύσουμε και μία πλατφόρμα διαφάνειας όπου οι κατάντι επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να επιδείξουν την, ε, τη δουλειά τους της δέουσας επιμέλειας. Γιατί κυρίες και κύριοι δεν υπάρχει κανένα καλύτερο απορριπαντικό από το φως του ηλίου, λέει ο μιλητής. Και με αυτόν τον τρόπο οι κατάντια επιχειρήσεις θα μπορέσουν και αυτές να συμμετάσχουν στην προσπάθεια που ήδη καταβάλουν οι εξαγωγείς. Οι εισαγωγείς. Και θα πρέπει και οι καταναλωτές και όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εμπόριο αυτό να βασιστούν σε μια σε σειρά κατευθύνσεων για την υπεύθυνη προμήθεια. Και έχουμε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή κάνει αυτή τη δουλειά στην Νότια Αφρική. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια συνολική προσέγγιση, ολοκληρωμένη προσέγγιση, γιατί είναι ένα περίπλοκο παζλ με πολλά επίπεδα και πολλά κομμάτια, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για μια αποτελεσματική υλοποίηση. Τώρα, για το νομοθέτημα που έχετε μπροστά σας, προτού σας πω τι κάνει, θα σας πω τι δεν κάνει. Δεν κάνει τα εξής. Δεν αλλάζει την ισορροπία που είχε επιτευχθεί στον κανονισμό ορυκτών εμπολέμων ζωνών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερον, δεν υπερβαίνει τα όρια της εξουσιοδότησης που μας παρέχεται. Θα θυμάστε ότι ο κανονισμός των ορυκτών εμπόλεμων ζωνών λέει ότι οι μελέτες ιδέους επιμέλειας θα μπορούν να υποβάλλονται προς έγκριση από την Κομισιόν και μετά θα πρέπει να έχουμε τη μεθοδολογία και τα κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των μελετών δέους επιμέλειας. Αυτό είναι που έχετε μπροστά σας, όπως ο εισηγητής ήδη σημείωσε. Εσύ έχεις αναμένο μικρόφωνο το Με μεγάλη χαρά λοιπόν να μοιραστούμε μαζί σας τα αποτελέσματα της ε, διάδρασης αυτής. Η κύρια προσέγγιση προς την εξουσιοδότηση είναι πολύ απλή. Έχουμε την πρόσθετη μεθοδολογία ε, που εγκρίθηκε από τον ΑΣΑ για τα συστήματα έγκρισης των ορυκτών, ώστε να έχουμε πλήρη έλεγχο του κεκτημένου μας, το οποίο είναι η αρχή που είχε αποτυπωθεί στον κανονισμό των ορυκτών εμπόλεμων ζωμών. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφή κριτήρια, όχι μόνο επιλεξιμότητας αλλά και αξιολόγησης. και για άλλες πηγές πληροφοριών όπως υπενόησε και ο εισηγητή. Δηλαδή για σκιώδεις ελέγχους. Και επ' αυτού προχωρούμε λοιπόν και υλοποιούμε. Ε, το άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η διαφάνεια. Έχουμε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, πολύ συγκεκριμένο καταμερισμό ευθυνών, καθηκόντων Συμμετοχή για, τους διάφορους, για τα διάφορα μέρη. Λαμβάνει υπόψη του επίση ότι εδώ είναι πολύ σημαντική η ανάλυση αυτή. Χρειάζεται ο χρόνος για να διατρέξουμε και να φτάσουμε στην κατάλληλη απόφαση για όλα αυτά τα προγράμματα δέους επιμέλειας. Και επομένω, δίνουμε στον εαυτό μας όχι πολύ χρόνο, αλλά το χρόνο που χρειάζεται. Εννέα μήνε. Και ένα-δύο ακόμα στοιχεία πρωτού ε, σας επιστρέψω το μικρόφωνο, Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι σε προηγούμενες συζητήσεις για τον κανονισμό αυτών κάποια σημεία ήταν πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο. Όλοι οι ενωσιακοί εισαγωγή θα πρέπει να συμμορφούνται, να έχουν όλα τα κριτήρια συμμόρφωση προς τις διατάξεις του κανονισμού, ανεξαρτήτως του κατά πόσον συμμετέχουν σε σύστημα συναλλαγής που έχει εγκριθεί από την Κομισιόν. Δεύτερον, η αξιολόγηση αυτών των συστημάτων συναλλαγών δεν θα μένουν μόνο στις πολιτικές και τα πρότυπα του, αλλά και στην υλοποίησή τους. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργούν και λειτουργούν σωστά. Να σας πω επίσης, μάλλον τέλος, ότι έχουμε υπογραμμίσει την σημασία της διαφάνειας σε όλη τη διαδικασία και να σας διατηρούμε ενήμερους για την υλοποίηση του κανονισμού και θα κλείσω χωρίς να πρωτοτυπήσω όπως και τα κράτη-μέλη εγκαίρως συνέταξαν τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες, θα ζητήσουμε και εμείς από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο να εξετάσει σύντομα, γρήγορα σας παρακαλούμε τον κατεξιό Η ιδάλω δεν θα μπορέσουμε να είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος για να υλοποιήσουμε το αντικείμενο του κανονισμού αυτού. Αυτά σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Ρινά. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Χαίρομαι διότι η Κομισιό έχει παρουσιάσει διάφορα σημεία θετικά. Δηλαδή πρώτα απ' όλα, και αυτό αποφαλούσε ένα ακρογωνιαίο λίθο του κανονισμού, για του οποίου είχαμε ερωτηματικά, το γεγονός ότι θα αναγνωρίζεται το, η μορφή της ε, ε, βιομηχανίας σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στον ΩΣΑ. Το θέμα αυτό της ευθυγράμμισης λοιπόν στις ισχύοντες κανόνες για το θέμα αυτό στον ΩΣΑ είναι ενθαρρυντικό. Δεύτερον, το γεγονός ότι όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτό το ειδικό σχήμα είναι ατομικά υπεύθυνε. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι χάνει κάθε επιχείρηση την ατομική της ευθύνη. Βλέπω λοιπόν ότι και πάλι αυτή την ευθύνη της κάθε επιχείρηση την έχει λάβει υπόψη η Επιτροπή. Τρίτο σημείο, το οποίο όμω δεν έχει εξηγηθεί με σαφήνεια από την Επιτροπή, αφορά την αξιολόγηση των πρακτικών των διαφόρων επιχειρήσεων. Είχαμε πει ότι θα μπορούσε να υπάρχει ε, και οικονομικός έλεγχος ε, σε κάποιες επιχειρήσεις με την βάση σφιγμομέτρησης που γίνεται βάση των ότι ισχύει για τι επιχειρήσει αυτέ, αλλά βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το λαμβάνει υπόψη. Διότι είδαμε ότι πάρα πολλέ φορέ υπήρχαν σκάνδαλα, ξέπλυμα χρήματο, διαφθορά. Στην και μετά είδαμε ότι υπάρχει πρόβλημα το 2016 τα θέματα του χρυσού. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχε η αναγνώριση ενός σχήματος που έπρεπε να ακολουθηθεί, υπήρχαν προβλήματα διαφοράς. διαφθοράς. Με συγχωρείτε. Και σήμερα αυτά τα οποία έχουμε βάσει των κανόνων της νομοθεσίας δεν μας προστατεύουν απολύτως. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν ποια είναι η θέση της σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εγγυηθεί το ότι τέτοιου είδους καταστάσεις θα μπορούσαμε να τις αποφύγουμε στο μέλλον. Επίσης, στα πλαίσια των κατεξουσιοδότηση πράξεων θα μπορούσε να γίνει ε, είπατε ότι θα, κατά περίοδους θα γίνεται αναθεώρηση. Θα μας πείτε ποια χρονική περίοδο θεωρείτε εσείς ως ε, περιοδικό έλεγχο. Εν, κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια. Ποια είναι η χρονική περίοδος στην οποία ορίζετε εσείς όταν μιλάτε για περιοδιωτικότητα. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να μιλήσω για την ε, περιδική αναθεώρηση. Το, το κόμμα μιλάει για αυτό το θέμα στον, στον αλλά δεν βλέπω αυτό να είναι κάτι το οποίο το εγκυάται η, ο κανονισμός κάτω κάτω εξουσιοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές στα πλαίσια αυτού του σχήματος υπάρχουν επιχειρήσεις που ε, ε, θεωρούνται χαμηλού κινδύνου, αλλά δεν είναι όλες έτσι. Πού λοιπόν υπάρχει η εγγύηση, ε, αναφέρομαι και πάλι στην εφοδιαστική αλυσίδα άρθρο 8, 4. Ε, Δεύτερη παρατήρηση. Τα ίδια αυτά τα σχήμα των βιομηχανιών, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΩΣΑ που χρησιμοποίησε και η Κομισιό, σύμφωνα με τη μεθοδολογία, πρέπει να ελέγχουν τα μέλη τους. Σε τακτά διαστήματα. Επίσης, για αυτό το θέμα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται. Θα πρέπει διάφορα ε, στοιχεία που αφορούν ότι έγινε τέτοιου είδου έλεγχος να μας παρουσιάζονται σε εμά. Επίσης, ο ορισμός που έδωσε ο ΣΟΣΑ για τον εφαρμογή. Και διαβάζω για την μεθοδολογία ευθυγράμμιση σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΣΑ. Σελίδα 6 λέγεται ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ορισμό που αφορά τα εκτήρια εφαρμογής από το πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μέτρων ώστε να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει πλήρη συμμόρφωση στα πλαίσια των επιχειρήσεων που συμμετέχουν εδώ. Πώς γίνεται αυτό, θα ήθελα να το καταλάβω καλύτερα. Κάτι άλλο. Ο κατάλογος όλων αυτών των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την δίξη και την επεξεργασία περαιτέρω αυτών των ορυκτών και μετάλλων. Γίνεται έλεγχος, αλλά δεν μπορεί να κάνει η αυτό τον έλεγχο. Τον κάνουν οι εθνικές αρχές. Αλλά Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε κάποιος να τον κάνει αυτό τον έλεγχο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις που υπάρχουν σε αυτόν τον κατάλογο πραγματικά ελέγχονται σωστά. Επίσης, κάτι άλλο που αφορά το δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι τα πήρατε όλα μαζί τα θέματα αυτά. Καταλαβαίνω ότι έχουμε δυσκολία με το να αποσαφινιστούν τα θέματα των εισαγωγών, διότι οι τελωνιακές αρχές δεν μας δίνουν εύκολα, δεν δίνουν εύκολα τα ονόματα των επιχειρήσεων αυτών στις ε, εθνικές αρχές. Δεδομένου ότι είναι εμπιστευτική κυρίως ε, η εισαγωγή χρυσού. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι έρχεται μια εθνική αρχή που είναι η τελωνιακή αρχή, που δεν δίδει τις απαραίτητες ε, πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι άλλες εθνικές αρχές ώστε να ελέγξουν τις περιχειρήσεις. Εκτός αν θέλουν να βγάλουν χρήματα από όλη αυτή την υπόθεση, αλλά εμείς δεν νομίζω ότι το θέλουμε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω πώς ε, διευθετείται αυτό το θέμα για τους πράσινους είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό πριν να μπορέσουμε να αποδεχθούμε το ότι ο κανονισμός αυτός κατά την μπορεί να γίνει αποδεκτός. Από εμάς ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Χέλμουτ Σόλτς μου ζήτησε να ε, συνεχίσω το διάλογο στο όνομα της GoNGL, αυτό κάνω λοιπόν. Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με την κατεύθυνση που έχουμε πάρει, έχουμε όμως κάποιες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η πρόταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιβολή του νόμου. Αυτό μπορούμε να το, να το κάνουμε ε, διευρύνοντας ε, τις διατάξεις του κανονισμού ώστε να καλύπτει όλες τις ε, επιχειρήσεις ε, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που διαθέτουν ε, στην αγορά τα προϊόντα αυτά. Επίσης μπορούμε να φροντίσουμε οι επιχειρήσεις να υποβάλουν πληροφορίες με εναρμονισμένο και διαφανή τρόπο και να φροντίσουμε η επικοινωνία των αρχών να βασίζεται στην καλή επικοινωνία και με ανοιχτά δεδομένα να έχουμε πλατφόρμα για ε, συχνούς ε, και τυποποιημένους ε, διαλόγους ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και να έχουμε διάταξη για τους αναφέροντες παρατυπίες, τους whistleblowers. Επίσης θα πρέπει να γίνονται έρευνες από τις αρχές της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, ναι, ε, έχω κάποια θέματα, έχω σημειώσει κάποια θέματα, αλλά οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο τα κάλυψαν όλα αυτά. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση και να προσθέσω μια παρατήρηση. Ε, καταρχάς, μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να αναφερθείτε στην δημιουργία επαφών παγκοσμίω όσον αφορά τις προσπάθειές μας. Τι γίνεται στην Κίνα, τι γίνεται στην Νότια Αμερική, αν γίνεται κάτι ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εάν γνωρίζουμε τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, θα ήταν χρήσιμο διότι έχουν και εκείνη συγκεκριμένο κανονισμό. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Η παρατήρησή μου ε, είναι να επαναλάβω αυτά που είπε ε, η τελευταία ομιλήτρια. Μιλήσαμε για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και όσον αφορά τα υλικά και όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Νομίζω όμως ότι αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι να επικεντρωθούμε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία, να επικεντρωθούμε στα ερωτήματα που ήδη έχουν τεθεί και φυσικά μετά την εφαρμογή του κανονισμού μας ε, το 2003, αν δεν κάνω λάθος, να έχουμε την πρώτη αναθεώρηση και τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, προ τη μία την άλλη κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σκέφτομαι το θέμα τη ε, διεύρυνσης τη πρόταση, διότι όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα χρειαζόμαστε ηλεκτρικούς συσσουρευτές, ηλεκτρικές μπαταρίες, όπου ε, περιλαμβάνεται και κοβάλτιο. Το 60% του κοβαλτίου προέρχεται από το Κονγκό. Και έτσι θα έχουμε σημαντική αύξηση των μπαταριών των συσσωρευτών στο μέλλον, εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας στον κανονισμό ε, του Δεκεμβρίου για το διοξίδιο του άνθρακα. Το κοβάλτιο, λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο ορυκτό που θα συμπεριληφθεί σε μια διεύρυνση της πρότασης αυτής. Αλλά βέβαια αυτό δεν αφορά την εφαρμογή της πρότασης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα το αποκαλούσα αυτό τσουνάμι ερωτήσεων. Συγχωρήστε μου αν στην προσπάθεια να επιπλέψω μου διαφύγει κάποια από τις παρατηρήσεις σας, αλλά είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω. Απαντήσεις και διαφαινήσεις. Τώρα, Κάποια από τα τελευταία σχόλια που έγιναν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει κανείς ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίηση των όσων έχουμε σήμερα. Δεν θα μπορέσουμε να τροποποιήσουμε το πλαίσιο αυτό μέσω του κατεξιότσιν κανονισμού. Οπωσδήποτε γνωρίζουμε τα θέματα, τις ανησυχίες δηλαδή που έχουν εκφραστεί για το πεδίο, όπως και των εμπορικών φορέων κατάντι. Όμως το νομικό μας πεδίο είναι ξεκάθαρα περιγεγραμμένο. Τώρα, λόγω αυτής της πλατφόρμας διαφάνειας, μεταξύ άλλων, θα δείτε ότι έχουμε προχωρήσει σε πολύ έντονη δραστηριότητα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια θετική προσέγγιση για αυτούς, για αυτές τις κατάντια επιχειρήσεις που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και που νομίζω ότι συνεχίζουν την όθηση που χρειάζεται ώστε οι περισσότερες όλες οι επιχειρήσεις να τηρούν τις δεσμεύσεις του πλαισίου αυτού. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσω ότι κοιτούμε και τις ε, συμφωνίες συναλλαγής αλλά και τον έλεγχό τους. Καταρχάς θα έχουμε πράγματι τους ε, λεγόμενους σκιώδεις ελέγχους. Για το πώς υλοποιείται το σύστημα συναλλαγών. Τα συστήματα αυτά επίσης θα τα αξιολογούμε αυτά, που είναι διαφορετικό από την αξιολόγηση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αυτά υπό το άρθρο 8.3 ε, του κανονισμού των ορεικτών εμπόλεμων ζωμών, που δεν μπορεί ο κατακυσότης να αλλάξει, αλλά και οι επιμέρους επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να και αυτές να αξιολογούν τη λειτουργία του. Και εδώ η λέξη κλειδί είναι η υπευθυνότητα Πρέπει λοιπόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις να τηρούν τις υποχρεώσεις και το πλαίσιο αυτό. Στον καταξιότητα κανονισμό επίσης θα βρείτε και νομίζω ότι εδώ απαντώ και στα απολύτως κατανοητά σχόλια που κάνατε. Τι γίνεται μετά αφού αξιολογήσουμε την ισοδυναμία όπως την ονομάζουμε ενός συστήματος συναλλαγής. Είναι σημαντικό να έχουμε σαφέστατες διατάξεις στην περίπτωση που εντοπίσουμε οποιαδήποτε απόκληση ή έλλειψη. Στο άρθρο 11 έχουμε μια σειρά από ισχυρές διατάξεις ώστε το συγκεκριμένο σύστημα να επιδιορθωθεί. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε ένα δυναμικό κανονισμό υπό τον οποίο όταν ένα σύστημα δεν τηρεί πλέον τις υποχρεώσεις του απορρίπτεται. Αποκλείεται. Για το θέμα της περιοδικότητας και του ελέγχου Έχουμε την γενική επανεξέταση που λαμβάνει η χώρα τακτικά. Η πρώτη θα είναι το 2023, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουμε συντάξει την κατεξότηση πράξη σημαίνει ότι έχουμε ενσωματώσει μία αρχή συνεχόμενης εξέτασης, λέει ο μιλητής. Δηλαδή, για οποιαδήποτε επιτυχή της δέωσης επιμέλειας καταβάλλεται μια συνεχή προσπάθεια εξέτασης και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σχετικά με οποιαδήποτε έλλειψη οποιοδήποτε επιμέρους συστήματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και γι' αυτό συμπεριλάβαμε συγκεκριμένα αριτά μια διάταξη στο 13.4 όπου Καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση του κανονισμού. Μέσω μιας τέτοιας ε, προσέγγισης θα μπορέσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση, εντάξει, να μην πω καθημερινά, αλλά σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο περιοδικότητας. για τις ε, πληροφορίες των τελωνιακών αρχών. Βεβαίως και θα έχουμε πρόσβαση σε αυτές και αυτό θα μας επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε και μια διάδραση ανταλλαγή με τους συναδέλφους των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε ζητήματα για οποιασδήποτε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και παρότι δεν ετέθη το ερώτημα αυτό από εσά. Να πω ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε αυτή την πληροφορία για διάφορα κατώτατα όρια που ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Έχουμε και το επίπεδο των κωδίκων TARIC 10 όπως ονομάζονται υποκώδικες τελωνιακούς που έχουν συλλεχθεί από τα κράτη-μέλη και που το τέλος του 2019 θα έχουμε επαρκή στοιχεία ώστε να εξετάσουμε τα όρια αυτά. Επίσης έχουμε πραγματοποιήσει μια προσπάθεια προσέγγισης πάρα πολύ σημαντική, πιο εντατική από ποτέ και ως τελευταία παραδείγματα να σας πω ότι ένα από τους συναδέλφου, ε, όπως έλεγα και πριν, είναι στην Νότια Αφρική για να ε, έχει επαφές με την ε, κοινότητα των εξορίξεων εκεί. Και στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου για τα υπεύθυνα ορυκτά στην Κολομβία πέρυσι ήμασταν ένας από τους συμμετέχοντες κλειδιά με ακροατήριο σημαντικές, σημαντικές επιχειρήσεις αμερικανικές και καναδικές που είναι κατάντι στο σύστημα αυτό και που είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, στο ανταλλακτήριο μεταλλευμάτων του Ντουμπάι και σε άλλα πολύ σημαντικά φόρα, όπου συμμετέχουν επιχειρήσεις που διαδραματίζουν ρολοκλειδί σε όλο αυτό το πλαίσιο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες προσέγγιση, outreach για να συνεννοούμεθα, είναι πολύ σημαντικές γιατί όπως θα γνωρίζετε ίσως και οι Κινέζοι αναπτύσσουν το δικό τους σύστημα, το δικό του πλαίσιο, το οποίο βέβαια, πώ να το πω, δεν παρέχει τη χρυσή ισορροπία και διαφάνεια παρέχει το δικό μας, και για τους Αμερικανούς ομολόγους μας είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια διότι τα πράγματα δεν κινούνται ακριβώς προς την ιδανικότερη των κατευθύνσεων. Με αυτά προσπάθησα να καλύψω τα πιο σημαντικά από αυτά που είπατε, από τις παρατηρήσεις σας. Ε, ίσως κάτι που δεν κάλυψα, ναι, ζητώ συγγνώμη, όταν γίνεται οποιαδήποτε ερώτηση είτε του Προέδρου είτε οποιοδήποτε μέλους πρέπει να απαντούμε. Αναφερθήκατε Πρόεδρε λοιπόν ιδιαίτερα στο θέμα του κουβαλτίου. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή καλύπτονται όλα τα ορεικτά που θα μπορούσαμε στα, στον κανονισμό για τα ορεικτά εμπολέμων ζωνών. Έχουμε ένα στρατηγικό ε, σχέδιο δράσεως για τις μπαταρίες, για τους σωρευτές από το 2016 και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε και πρωτοβουλίες ε, του κλάδου που θα μπορούσαν να ανακύψουν, να αναδυθούν. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε ακριβώς καλύψει το 100% των πάντων, αλλά όλα βρίσκονται στις κεραίες του ραντάρ μας. Εξού και το σχέδιο του κατεξιότητας κανονισμού που έχετε μπροστά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Μία παρατήρηση πάντα συμβαίνει, όχι μόνο σε αυτή την νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα παίζει σημαντικό ρόλο. Γιούντιθ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με επιτρέπετε να επανέλθω. Ε, δεν είμαι βέβαιη ότι κατάλαβα την απάντησή σας. Καταρχάς, όσον αφορά την περιοδική επανεξέταση, μας εξηγήσατε ότι υπάρχουν δυνατότητες στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Άλλοι να ε, το επισημάνουν εάν θεωρούν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα καλά. Πολύ ωραίο αυτό. Αναφερθήκατε στο άρθρο 13.4 που δίνει τη δυνατότητα αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωραία αλλά αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε μηνύματα απ' έξω. Και αυτό ε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο με το να ε, τηρούμε τον, ε, το άρθρο 8.4 του ε, κανονισμού που λέει ότι πρέπει να ενσωματώσουμε την περιοδική αναθεώρηση. Πού υπάρχει αυτό στην κατεξοδότηση πράξη. Ε, ευχαρίστω θα λάβω την απάντηση γραπτό, διότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η άλλη μου παρατήρηση έχει να κάνει με τη συνεργασία ανάμεσα στι τελωνιακέ αρχέ και την Εθνική Αρχή. Εσεί εξηγήσατε ότι ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχετε πρόσβαση σε τέτοιε πληροφορίε. Αλλά αυτό δεν απαντά στη δική μου ερώτηση. Ξεκινήσατε την ε, παρουσίασή σας αναφερόμενος στο, στον ήλιο που είναι ε, το καλύτερο απολυμαντικό. Ε, χρειάζεται όμως να δημοσιεύουμε τους εισαγωγείς ε, από ε, εμπόλεμες ζώνες. Ε, εάν όμως δεν διατίθενται οι πληροφορίες αυτές, ε, η κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να διπλοτσεκάρει τι ακριβώς γίνεται. Το θέμα της δέουσας επιμέλειας συνδέεται στενά με την διαφάνεια. Πρόεδρος, δύο ερωτήσεις, δύο σύντομες απαντήσεις θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτησή σας. Αυτό που προσπάθησα να εξηγήσω είναι ότι οι προσδοκίες μας είναι ότι θα έχουμε πολλές πληροφορίες που θα έρθουν όχι μόνο από εσά, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται, χάρη στην πλατφόρμα της ε, διαφάνειας, αλλά και στα πλαίσια του όσα έχουμε την δυνατότητα να εντοπίσουμε τα θέματα για τα οποία υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος στο πλαίσιο αυτής της δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να πω και η συνάδελφος μου λέει ότι μπορώ να σας δώσω και κάποιες άλλες πληροφορίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην παράγραφο 12 φερρυπίν θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε το ότι έχουμε έγκαιρα δημόσια ενημέρωση. Όταν αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί βεβαίω. Και χάρη στους διάφορους μηχανισμούς που έχουμε στον κανονισμό, μπορούμε να έχουμε διάφορα στοιχεία που μας επιτρέπουν να ενεργήσουμε αμέσως. Και αυτό είναι κάτι βάσει του 8.4 όπως είπατε. Και βάση περιπτώσει τι θα γίνεται και τακτική αναθεώρηση και εποπτεία. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Τη δεύτερη τώρα. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Είναι σημαντικό για μας να έχουμε τις προφορίες που μας επιτρέπουν να ενεργήσουμε. Και αυτό είναι το καλύτερο καθαριστικό, όπως σας είπα. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι, το, οι κανόνες του απορρίτου θα τηρούνται απολύτως, δεν θα υπάρχουν αποκλήσεις, ώστε να δούμε αν υπάρχουν παραβιάσεις σχέση με την τελωνιακή νομοθεσία. Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών θεμάτων, έχοντας πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες κάθε επιχειρήσεις χωριστά, χωρίς να παραβιάζουμε τις διατάξεις που αφορούν την τελωνιακή νομοθεσία. Και εσείς και οποιοδήποτε άλλο θέλει να κάνει το έλεγχο μπορεί να μας ζητήσει οτιδήποτε στα πλαίσια αυτών των διατάξεων. Βεβαίως. Πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και δυνατοί για να προχωρήσουμε, αλλά πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Οι συντονιστές θα αποφασίσουν μέσα στο Φεβρουάριο ποια θα είναι η περίοδος εποπτείας ελέγχου Ελπίζουμε ότι και το Μάρτιο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ολοκληρώθηκαν τα σημεία 11 και 12. Το 13 στα διάφορα. Δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Και 14. Επόμενη συνεδρίαση 18 και 19 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.